Ευχαριστώ κύριε Σένκοβιτς. Σας ευχαριστώ γιατί δείξατε και τις γλωσσικές σας ικανότητες χρησιμοποιώντας πολλές γλώσσες και χαίρομαι και για το γεγονό ότι χρησιμοποίησατε και τη μητρική μου γλώσσα τα γερμανικά. Έρχομαι τώρα στους συντονιστε. Ο κύριος Βιμ Βαντενκάμπ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Δεν μιλάτε ακόμα Ολλανδικά, αλλά νομίζω ότι κάτι θα κάνουμε για αυτό το θέμα. Σας καλωσορίζω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εξ ονόματος της του ΕΛΚ. Θα θέλαμε να συνεργαστούμε μαζί σας με ένα φιλόδοξο και δίκαιο τρόπο. Χωρίς τις μεταφορές όλα είναι στατικά. Φυσικά ακόμα και η, Ευρώπη, η ευρωπαϊκή ιδέα. Έχω ορισμένα ερωτήματα. Καταρχήν, η λευκή βίβλος για τον οδικό χάρτη για μια ενιαία ζώνη μεταφορών στην Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει θέσει ορισμένε προτεραιότητε, τι οποίε τι αποδέχεστε εσεί ή όχι. Θέλετε να τι αλλάξετε, ποια είναι τα σχέδιά σα για το θέμα αυτό. Δεύτερο ερώτημα. Η χρηματοδότηση των σχεδίων TNT, το αναφέρατε αυτό. Μιλάτε για 300 εκατομμύρια, δισεκατομμύρια από τον κύριο Γιούνκερ που έχουν αναγγέλθει Πόσα από αυτά τα 300 δισεκατομμύρια όμως θα αφιερωθούν στα προγράμματα και τα σχέδια του TNT. Θα θέλαμε να έχουμε κάποια πιο συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία. Και τέλος ένα πιο δύσκολο σημείο. Η συνεργασία με τους άλλους επιτρόπους και τους άλλους γενικούς διευθυντές. Έχουμε σημειώσει ότι ο Επίτροπος Μεταφορών βρίσκεται πολλές φορές σε αντιπαράθεση με τον Επίτροπο Ανταγωνισμού, τον Επίτροπο ε, <clears throat> Περιβάλλοντος κτλ. Πώς θα αντιμετωπίσετε λοιπόν ένα τέτοιο πρόβλημα, γιατί οι μεταφορές πρέπει να παίξουν ένα προεξέρχοντα ε, ρόλο στην κοινωνία μας. Και τέλος, επειδή έχω λίγα δευτερόλεπτα ακόμα, θα ήθελα να σας, πω, να σας ρωτήσω τι θα κάνετε για αυτούς που έχουν περιορισμένη κινητικότητα. Μιλήσαμε για αεροπλάνα, για τρένα, για μεγάλα σχέδια. Τι θα κάνετε όμως για τα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. Θα κλείσω εδώ, δεν ήθελα να ε, πάω πολύ γρήγορα και σας ευχαριστώ. Έχετε το λόγο. Θα βελτιώσω τα Ολλανδικά μου, σας το υπόσχομαι. Για να έρθω στα ερωτήματά σας. Όταν συζητούσα με τους συναδέλφους μου στην Κομισιόν, με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να καθορίσουμε τον οδικό χάρτη για τα επόμενα πέντε χρόνια, το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξα είναι ότι όσο πιο σύντομα έρθει η μεταρρύθμιση της Λευκής Βίβλου, τόσο και καλύτερα. Γιατί πιστεύω ότι το δίδαγμα των τελευταίων ετών ήταν ότι ήταν κάπως καθυστερημένα η Λευκή Βίβλος στην προηγούμενη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και φυσικά έπρεπε να τροποποιηθούν τα σχέδια για νομοθεσία. Σας υπόσχομαι λοιπόν θα κάνω ό,τι μπορώ για να μπορέσω να επιταχύνω τη διαδικασία μεταρρύθμισης της Λευκής Βίβλου. Μέχρι τώρα μπορούμε να πούμε σίγουρα ότι η πρόοδος για το σχέδιο αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντική. 24 από 40 δράσεις που προβλεπόταν στη Λευκή Βίβλο έχουν ήδη ή περατωθεί ή ξεκινήσει. Και φυσικά είμαι έτοιμος να τα συζητήσω και με τους συναδέλφους μου στην Κομισιόν, γιατί αυτό είναι ένα έγγραφο το οποίο πρέπει να υποστηριχθεί από το σύνολο της Επιτροπής και μετά θα επανέλθει σε εσά και θα σας ζητήσει η Κομισιόν να το επεξεργαστείτε μαζί μας. Για τα σχέδια TNT και τα 300 δισεκατομμύρια, τι επενδύσει των 300 δισεκατομμύρια. Ξέρετε ότι 26 δισεκατομμύρια για τα σχέδια TNT είναι πολλά λεφτά, αλλά είναι μια σταγόνα εν το ωκεανό. Αν δείτε τι χρειάζεται η Ευρώπη, χρειαζόμαστε πολύ μεγαλύτερη χρηματοδότηση. Πιστεύω ότι καλά σχέδια υποδομών, σχέδια που ευνοούν την μελλοντική ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων είναι σχέδια όπου μπορούν να υπάρχουν και πολλές προοπτικές για επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα. Μπορούμε λοιπόν να προωθήσουμε αυτή την εταιρική σχέση δημόσιου ιδιωτικού τομέα και να έχουμε πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει επιτευχθεί και χάσει τη δική σας συμβολή μέσα στις ε, νέες δημοσιονομικές προοδίκες Ακριβώς πώς θα γίνει αυτό και πόσο ποσοστό αυτό το κονδυλίων θα πάνε στη δημιουργία υποδομών είναι δύσκολο να σας το πω τώρα, αλλά είναι δύσκολο να βρούμε εξίσου ελκυστικά σχέδια για εταιρική σχέση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και για το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που ε, επιτυγχάνει αυτή η εταιρική σχέση. Φυσικά θα πρέπει να υπάρξει και συνεργασία με όλους τους ε, συναδέλφους στην Κομισιόν και τους αντιπροέδρους και οι ανάδρομες ροές ε, και αυτές είναι στοιχεία τα οποία θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Η κυρία Τίσεν θα δώσει μια απάντηση πιστεύω για τα θέματα προσβασιμότητας που περιλαμβάνει και τα προβλήματα των ανθρώπων με περιορισμένη κινητικότητα. Σας ευχαριστώ για την τήρηση του χρόνου και περνάμε στον επόμενο μιλητή, ξενόμα της Σοσιαλιστικής Ομάδος τον κύριο Ερτούχ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κάθε επιτυχία από τη Σοσιαλιστική Ομάδα. Έρχομαι στο πρώτο μου ερώτημα τώρα που έχει να κάνει με το κοινωνικό δίκαιο και τα θέματα της εφαρμογής του. Τις κοινωνικές πτυχές τις θεωρούμε ότι είναι ένα σημαντικό στοιχείο της ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί. Θα ήθελα να ξέρω αν συμφωνείτε ότι η διατήρηση των κοινωνικών δικαιωμάτων θα πρέπει να διατηρηθεί σε όλο το χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν συμφωνείτε αν θέλετε πράγματι να τα εφαρμόσετε και στην πράξη. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι το θέμα της λεγόμενης βιώσιμης κινητικότητας της πόλης. <clears throat> Βλέπουμε ότι στις πόλεις υπάρχει όλο και μεγαλύτερη πίεση για τις μεταφορές και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Πώς ε, ε τοποθετήστε σε σχέση με την ε, τωρινή πολιτική κινητικότητα της πόλης που βλέπετε σφάλματα και που θεωρείτε πρέπει να υπάρξουν τροποποίησεις ο διαμερισ... η, το... Ε, από κοινού χρήση αυτοκίνητων παραδείγματος είναι ένας σημαντικός ε, χώρος. Ε, μπορεί η Κομισιόν να ζητήσει από τα κράτη-μέλη να επενδύσουν περισσότερο στο τομέα αυτό και στην δημόσια, δημόσιες μεταφορές και όχι μόνο στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα τρίτο στοιχείο έχει να κάνει με τις λιμενικές, τα λιμενικά θέματα. Το πακέτο για την πρόσβαση στα λιμάνια και την ε, διαφάνεια σε σχέση με τη χρηματοδότηση είναι πολύ σημαντικό και αυτό συνάπτεται με τις κρατικές επιδοτήσεις. Πώς θα αντιμετωπίσετε εσείς τις προσπάθειες για να υπάρχουν σαφείς κανόνες για τις υποστηρίξεις και πώς θα εξασφαλίσετε ότι αυτές οι ρυθμίσεις δεν θα αναχαιτιστούν από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Και έρχομαι τώρα στα λεγόμενα μεγάλα ε, για τα ε, μεγάλα πλοία και επίσης αν θα μπορέσει η Κομισιόν να προωθήσει νέα νομοθεσία για, την, ε, το συνδρομικό κλάδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Κύριε Θα προσπαθήσω να απαντήσω τηλεγραφικά γιατί θέσατε πάρα πολλά θέματα ταυτόχρονα. Καταρχά σχετικά με τα κοινωνικά δικαιώματα και τις κοινωνικές κατακτήσεις νομίζω ότι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα πράγμα ισχύει. Όταν προετοιμάζουμε τις νομοθετικές προτάσεις και όταν τις βάζουμε σε αξιολόγηση για τη μελέτη των επιπτώσεων το ερώτημα το οποίο πρώτα θα τίθεται είναι το πώς αυτό θα επηρεάσει την απασχόληση στην Ευρώπη. Θα δημιουργήσουμε νέες θέσεις απασχόλησης ή θα δημιουργούμε προβλήματα ε, στους εργαζομένους. Νομίζω ότι αυτή είναι η βασική αρχή την οποία πρέπει να σεβαστούμε και στον τομέα των μεταφορών. Για να είμαι ειλικρινής και βλέποντας το τι συνέβη τα τελευταία χρόνια θα μπορούσαν τα πράγματα να πάνε καλύτερα σε σχέση με τον κοινωνικό διάλογο. Γνωρίζω ότι διεξάγεται ο κοινωνικός διάλογος. Γνωρίζω ότι κυρίως οι συζητήσεις γίνονται σε τεχνικό επίπεδο και για να δημιουργηθεί ε, αν θέλετε περισσότερο ένα καλύτερο κλίμα εμπιστοσύνης απαιτείται περισσότερη συνεργασία ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους. Τώρα για τις λιμενικές εγκαταστάσεις και τους λιμένες γενικά. Αυτό είναι ένας τομέας στον οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε με μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Έχουμε αφήσει πίσω μας δύσκολες στιγμές. Υπάρχει τώρα πλέον μια τρίτη πρόταση για τις λιμενικές εγκαταστάσεις. Θα συνεργαστώ μαζί σας και με τους κοινωνικούς εταίρους για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα των λιμένων. Γιατί είναι πραγματικά οι θύρες της Ευρώπης και απαιτείται να τις συνδέσουμε με τα TEN, με τα διευρωπαϊκά δίκτυα και όχι μόνο σε σχέση με τους τρεις λιμένες στους οποίους αναφέρθηκα ήδη, αλλά το σύνολο των λιμενικών εγκαταστάσεων. Τώρα, για την αηφορία στις αστικές μετακινήσεις. Η πλειοψηφία των Ευρωπαίων ζουν στις πόλεις και τα περισσότερα ατυχήματα ε, γίνονται στην πόλη, οι εκπομπές είναι περισσότερες ε, στις πόλεις. <clears throat> Είναι λογικό λοιπόν να υπάρξουν ισχυρές πολιτικές για τις πόλεις. Δυστυχώς όμως αυτό δεν το συμμερίζονται ε, πολλές χώρες μέλη. Υπάρχουν τα θέματα της επικουρικότητας εδώ και θα πρέπει να τα συζητήσουμε μαζί τους. Όταν δείτε πώς οι δήμαρχοι βλέπουν το θέμα, πιστεύουν οι δήμαρχοι ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ευρωπαϊκή αντιμετώπιση, να υπάρξει μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα αστικής κινητικότητας μέσω συγκεκριμένων προγραμμάτων για να μπορέσουμε να ε, μοιραστούμε τις γνώσεις μας, τις βέλτιστες πρακτικές προς το καλό των πολιτών και το καλό του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ. Ζήλε, σας ευχαριστώ για την εισαγωγή σας κύριε Σεύκοβιτς. Από πλευράς της πολιτικής μας ομάδας θα θέλαμε να έχουμε μια σωστή συνεργασία μαζί σας. Ένα θέμα το οποίο θα ήθελα να θέσω. Εμείς εδώ στην Επιτροπή μας έχουμε ε, ανησυχίες για τους λεγόμενους διαδρόμους του Connecting Europe ε, επίσης η συμμετοχή κοινοτική σε τέτοια προγράμματα είναι ιδιαίτερα υψηλή. Ε, οι κανόνες λένε ότι μέχρι το τέλος του 2016, εφόσον δεν συνεχιστούν ορισμένα προγράμματα, θα πρέπει να εφαρμόσει την αρχή του ε, χρησιμοποίησε τις πιστώσεις ή χάσε τις πιστώσεις. Οπότε τι θα κάνετε. Πολλές αποφάσεις μερικές φορές εφαρμόζονται μόνο σε μία χώρα μέλος ε, κάτι το οποίο φυσικά δεν ε, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αντιπροσωπευτικότητα των προγραμμάτων αυτών. Το Connecting Europe λοιπόν θα πρέπει να αφορά πολλές χώρες κάθε φορά. Τώρα, οι υπερτήσει στην πολιτική αεροπορία. Στα πλαίσια της κρίσης με την ε, Ρωσία κάποιες, ε, κάποια Ευρωπαίοι αερομεταφορείς δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν την, ε, τον, σι, τον σιβηρικό εναέριο χώρο, λέει ο ομιλητής. Λοιπόν, η Ρωσία εδώ θα πρέπει ε, να σταματήσει ίσως να εισπράττει χρήματα από τους Ευρωπαίους αερομεταφορείς σε αυτή την περίπτωση. τι μέτρα, τι αντίμετρα θα έλεγα καλύτερα σκοπεύετε να λάβετε εις βάρος της Ρωσίας γύρω από την υπόθεση αυτή. Σας ευχαριστώ κύριε Ζήλε για τις δύο ερωτήσεις σας. Ξεκινώντας με τους διαδρόμους του Connecting Europe. Υπάρχουν κάποια προβλήματα σε πολλές περιπτώσεις, διαπιστώνονται ιδιαίτερα στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη σχετικά με την δυνατότητα απορρόφησης των πιστώσεων. Είναι αλήθεια ότι το 2016 θα είναι μια κρίσιμη χρονικά στιγμή και θα πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί και να δείξουμε ότι ε, ε, το εννοούμε αυτό το οποίο λέμε. Εάν φανεί ότι ε, δεν έχουν σεβαστεί κάποιοι εμπλεκόμενοι ε, τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει, τότε το θέμα της χρηματοδότησης με κάποιο τρόπο θα πρέπει να τεθεί. Ήδη έχουμε περάσει σε διαφορετικό πλέον πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και θα έπρεπε να έχουν γίνει εν τω μεταξύ όλες οι αλλαγές που θα διασφαλίσουν την αύξηση της απορροφητικότητας από τα κράτη-μέλη και ε, θα πρέπει να εφαρμοστεί η αρχή use it or lose it. Ε, βέβαια πρέπει να είμαστε δίκαιοι απέναντι στα κρατημέλη γιατί μερικές φορές είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει κανείς να ε, εφαρμόσει όλα αυτά τα προγράμματα. Γι' αυτό λοιπόν θα τα εξετάσουμε αυτά προσεκτικά και θα τους δώσουμε με δίκαιο τρόπο μια προειδοποίηση. Κοιτάξτε, αν δεν τα χρησιμοποιήσετε τώρα κινδυνεύετε να τα χάσετε. Όλοι ελέγχουν εδώ και οι ελεγχόμενοι είναι αυτοί και ελέγχοντες είμαστε εμείς αλλά και εσείς σαν κοινοβούλιο. Πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί λοιπόν σε σχέση με όλα αυτά και νομίζω ότι με την στήριξή σας θα τα λύσουμε τα προβλήματα. Τώρα για την υπέρπτυση στη Σιβηρία. Ξέρετε ότι οι σχέσεις μας με την Ρωσία είναι ιδιαίτερως περίπλοκες, όχι μόνο στον πολιτικό τομέα, αλλά και στον τομέα των οικονομικών και τις μεταφορές. Θα σταθώ στο θέμα των υπερπτήσεων. Είναι ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζουμε για πάρα πολλά χρόνια. Είχαμε πάρει πάρα πολλές υποσχέσεις. Η τελευταία υπόσχεση των Ρώσων είναι ότι εφόσον μπούμε στον ΠΟΕ θα καταργήσουμε τα τέλη αυτά, τη τέλη υπέρπτυσης και δεν θα τα χρεώνουμε πλέον. Ε, μέχρι τώρα όμως οι Ευρωπαίοι αερομεταφορείς πληρώνουν πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ τα οποία χρησιμοποιούνται ουσιαστικά σαν επιδότηση ε, των ρωσικών αερογραμμών οι οποίες εταιρείε οι ρωσικές κάνουν τα ίδια δρομολόγια με τις δικές μας. Αυτά δεν είναι σωστά πράγματα. Κανονικά θα έπρεπε να εξομαλυνθούν οι σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία. Αυτό ελπίζω και θα εργαστώ γι' αυτό. Είμαι πεπισμένος ότι μπορούμε να πείσουμε τα κράτη-μέλη ότι θα πρέπει ε, καλό να είναι οι Ευρωπαίοι να έχουν μία φωνή απέναντι στη ρωσική πολιτική και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πιέσει να υπάρξει μια συμφωνία για την υπέρκτηση της Σιβηρίας γιατί τα τέλη τα οποία ε, εισπράττουν είναι κάτι το οποίο δεν είναι συμβατό με τους διεθνείς κανόνες. Ευχαριστώ κύριε. Η κυρία από την ομάδα των φιλελευθέρων καλώ ήρθατε κύριε υποψήφια. Περιμένω τις απαντήσεις σας για τις ερωτήσεις που θα σας διατυπώσω. Θα ήθελα να επικεντρωθώ όπως και εσείς στο μεγαλύτερο μέρος στην αρχή της εκθέσης στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο των μεταφορών που βεβαίως και όλοι επιθυμούμε και ιδιαίτερα θα ήθελα να βάλω έμφαση στο χώρο των θαλασσίων μεταφορών. Αναφερθήκατε στη σημασία των λιμένων και ιδιαίτερο αυτό που με ικανοποίησε ήταν αυτό το οποίο ε, αναφέρατε για τις εσωτερικές πρώτες οδούς και τη σημασία τους που μπορούν να σημάνουν και αποσυμφόρηση των οδικών μεταφορών και την ενίσχυση βέβαια των θαλασσιών μεταφορών. Αυτό πρέπει να μπει μέσα στι θαλασσιέ μεταφορέ, γιατί έχουμε συζητήσει για ένα ε, δίκτυο των συντηροδρόμων. Πρέπει να κοιτάξουμε και τι θαλάσσιε μεταφορέ και κυρίω τι εσωτερικέ πλωτέ οδού, όπου μα είπατε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο δυναμικό ακόμα που δεν έχει αξιοποιηθεί. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να ρωτήσω το εξή θα πρέπει να αναπτυχθούν, δηλαδή να, βάλουμε πιο, να χτίσουμε πιο ψηλές γέφυρες, να σκάψουμε, να ανοίξουμε όχθες ε, σε ορισμένες περιοχές όπως και στην ιδιαίτερη μου πατρίδα. Αυτό πώς νομίζετε ότι μπορεί να γίνει, γιατί υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες κατά την υλοποίηση, επί παραδείγματι... Το ζήτημα της ε, αντιδράσεως πολιτών ως προς την ε, διάνοιξη ε, πλωτών οδών στον Δούναβη ή στον Έλβα ακόμα έχουμε ε, δυσκολίες συνεργασίας μεταξύ Τσεχίας και Γερμανίας. Πώς μπορείτε λοιπόν να ε, οθήσετε τα κράτη-μέλη σε μια πιο καλή συνεργασία στον τομέα αυτών. Παρακαλώ, απάντηση. Χωρίς μικρόφωνο. Ναι, ευχαριστώ κυρία Μάισνερ για την ερώτησή σας. Έχετε πολύ το δίκαιο ότι δυστυχώς οι εσωτερικές πλωτές οδοί και οι μεταφορές αυτές έχουν παραμεληθεί κάπως. Και λόγος ήταν ότι ο στόλος ήταν παλαιωμένος, απαρχαιωμένος, δεν είχαν σωστή συντήρηση, εσωτερικές πλωτές οδοί και ότι ήταν πολύ κατακαιρματισμένος ο κλάδος, κυρίως με πολύ μικρές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οικογενειακές ακόμη μικροεπιχειρήσεις οι οποίες ε, δυνατούν να κάνουν πραγματικά μεγάλες επενδύσεις και να βοηθήσουν έτσι στην ε, μεγέθυνση του κλάδου πέρα από αυτή την πολύ περιορισμένη κλίμακα. Γι' αυτό λοιπόν με χαρά βλέπω τα όσα έχουν γίνει και πιστεύω ότι μπορούν να βοηθήσουν πολλά στην τόσο υποσχόμενη αυτή ε, βιομηχανία, στον κλάδο αυτόν τον τόσο υποσχόμενο και οικολογικά αν δει κανεί δηλαδή πόσα μεταφορά μπορούμε να φορτώσουμε πάνω σε μια μαούνα ή τι είδου εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα μπορεί να έχει σε σχέση με άλλων τύπων μεταφορέ, αλλά και τι είδου δυνατότητες προσφορά ε, διασυνδέσεων μεταξύ λιμένων μπορεί να σημάνουν αυτές οι εσωτερικέ πλωτέ οδοί, βλέπουμε ότι έχει τεράστιο δυναμικό αυτό ο κλάδο. Εάν λοιπόν με στηρίξετε και με βοηθήσετε στην υπόθεση αυτή, εγώ θα ήθελα να αξιοποιήσω το πρόγραμμα Ναϊάδες ώστε να βοηθήσω στην ανοικοδόμηση του κλάδου των εσωτερικών πλωτών οδών, ε, να βοηθήσω στην ανακαίνιση του κλάδου των πλοίων, στον ανασχεδιασμό κατά τρόπο οικολογικό και σύγχρονο των πλωτών οδών, κατά τρόπον ώστε να ανταποκρίνονται σε όλες τις απαιτήσει μιας σύγχρονης μορφής εσωτερικών πλωτών μεταφορών. Και βεβαίως θα χρειαστεί και η στήριξη και η εντατική συνεργασία των κρατών μελών για την διατήρηση ενός υψηλού επίπεδου πλοηγημότητας ε, στις εσωτερικές πλωτές οδούς. Ξέρετε ότι η πατρίδα μου, ιδιαίτερη η Μπρατισλάβα, πάνω στο Δούναβι, μου επιτρέπει να γνωρίζω πολύ καλά τι είδους προβλήματα μπορεί να υπάρχουν και σε σχέση με τα γειτονικά κράτη. Ε, χρειάζεται λοιπόν πρόοδος είπα, στο τομέα αυτόν. Με ενθαρρύνει ιδιαίτερα το γεγονός ότι η πλογιμότητα του ε, Δούναβι έλαβε ιδιαίτερη σημασία στην ε, τοποθέτηση των κρατών της στρατηγικής για το Δούναβι έδωσε έτερη έμφαση, είπαν ότι υπάρχει δυναμικό, θέλουν να δώσουν νέες δυνατότητες και στην περιφέρεια και στις σταστικά κέντρα και τις μικρότερες πόλεις που βρίσκονται πάνω στον Δούναβι και πιστεύω ότι θα μπορούσαμε έτσι να καθησυχάσουμε και τους πολίτες ως προς τα προβλήματα που τους απασχολούν, δίνοντάς τους ότι υπάρχει δυναμικό, ένα δυναμικό το οποίο μπορούμε αναζωογονώντας αυτές τις οδούς, και αυτόν τον τρόπο μεταφοράς να στηρίξουμε και να βοηθήσουμε ιδιαίτερα και τις περιφέρειες και τις πόλεις. Είμαι πεπισμένος ότι αυτό είναι κάτι που μπορούμε και πρέπει να πράξουμε. Ευχαριστώ. Μαρία Κίλαρ. Κυρία Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήλθατε. Κύριε Θα έχω να σας θέσω τρία ερωτήματα. Πρώτον για τις συνθήκες εργασίας. Όταν έχουμε όλο και μεγαλύτερο παγκόσμιο ανταγωνισμό, υπάρχει όλο και μεγαλύτερη πίεση στις αγορές μεταφορών και φαίνεται ότι οι θέσεις εργασίας στον τομέα των μεταφορών κινδυνεύουν να μειωθούν κάτι το οποίο θα θίξει την βιώσιμη και ασφαλή κινητικότητα. Πώς θα εξασφαλίσετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα επιταχύνει την υποβάθμιση της ευρωπαϊκής πείρας γνώσης και πείρας και την ύπαρξη <clears throat> εργαζόμενων στον τομέα μεταφορών που έχουν αφοσίωση στον τομέα αυτό. Ιδίως στην ε, αεροπορία οι λεγόμενες εταιρείε χαμηλού κόστους παίζουν κορώνα γράμματα την ασφάλεια και εφαρμόζουν συνθήκες εργασίας όλο και χειρότερες. Είναι έτοιμη η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει τι ασφαλείς συνθήκε εργασία και ένα τρόπο εργασίας που αποτρέπει το κοινωνικό dumping. Ποια είναι τα σχέδιά σας επίσης για τους στόχους εκπομπών και ε, ψηφιακή ατζέντα. Πώς θα εξασφαλίσουμε την ε, οικονομική ανάκαμψη στον τομέα των μεταφορών και, θα μπορέ, και πώς θα μπορέσουμε να προωθήσουμε την ε, ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και την ευμάρεια των πολιτών της. Η ψηφιοποίηση, η ψηφιακή ατζέντα είναι πάρα πολύ σημαντική για τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις και βοηθάει και σε θέματα κινητικότητας και σε λύσεις προβλημάτων επιμελητίας. Είναι όμως ακόμα στα γενοφάσκια της αυτή η διαδικασία στον τομέα μεταφορών, αλλά πιστεύουμε ότι χάρη στην ε, χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών θα ανοίξουν πολλές δυνατότητες. Φαίνεται όμως ότι οι ανταγωνιστές μας, οι ΗΠΑ, η Κίνα και άλλες χώρες χρησιμοποιούν περισσότερο τις ψηφιακές δυνατότητες από εμά. Ελπίζω θα μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε και εμείς στην ξηρά, στη θάλασσα και στον αέρα, να δώσουμε περισσότερες δυνατότητες στα λιμάνια, τα αεροδρόμια και στους σιδηροδρόμους χωρίς κοινωνικό ντάμπινγκ. Πώς θα προωθήσετε λοιπόν τον τομέα μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να χρησιμοποιήσει περισσότερο τις ψηφιακές τεχνολογίες για να γίνει και πρωτοπόρος ο τομέας αυτός σε ό,τι αφορά την δημιουργία ενός διαλειτουργικού και βιώσιμου χώρου μεταφορών. Κύριε υποψήφιε επίτροπε, έχετε το λόγο, αλλά πρέπει να λάβετε υπόψη και το χρόνο γιατί το ερώτημα ήταν πράγματι μακροσκελές. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, <clears throat> συμμερίζομαι αυτά τα οποία είπε η αξιότιμη βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν δείτε τους ε, οδηγούς θα χρειαστούμε χιλιάδες οδηγούς επιπλέον στην Γερμανία και στην Ολλανδία. Βλέπετε ότι πάρα πολλοί από τους ε, μηχανοδηγούς των τρένων θα αποσυρθούν, θα πάρουν σύνταξη και θα χάσουμε την μεγάλη τους γνώση. Έχουμε χιλιάδες ναύτες από τις Φιλιππίνες στην ναυτιλία μας γιατί δεν μπορούμε να δώσουμε κίντρα στην ε, νέα γενιά που είναι η πιο άνεργη νέα γενιά μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο να πάρει αυτές τις θέσεις εργασίας και να εργαστεί στον ε, ναυτιλιακό τομέα, στις μεταφορές. Το πρώτο πράγμα λοιπόν το οποίο χρειάζεται είναι να αλλάξουμε την αντίληψη που έχουμε για τις μεταφορές. Θα πρέπει να εξηγήσουμε καλύτερα και να παρουσιάσουμε τον τομέα αυτό σαν ένα εργαλείο εξυγχρονισμού, σαν ένα οικονομικό κλάδος όπου μπορεί πράγματι κανείς να χρησιμοποιήσει υψηλές τεχνολογίες. Ένα τομέα όπου υπάρχει μια βιομηχανία που προετοιμάζει το μέλλον. Και αυτό πρέπει να γίνει γνωστό και στα σχολεία. Θα πρέπει να εργαστούμε και με τους κοινωνικούς εταίρους σε διάφορα επίπεδα για να βελτιώσουμε τις συνδίκε εργασίας. Γιατί πολλές φορές αυτό είναι το πιο σημαντικό κίνητρο. Τι είδους ε, κοινωνικές συνθήκες εργασίας, τι είδους ε, αποδοχές θα έχει κάποιος ο οποίος θέλει να εργαστεί στον τομέα μεταφορών. Εάν θέλουμε να είναι ελκυστικό ο τομέας για να αντικαταστήσει αυτούς οι οποίοι θα ε, συνταξιοδοτηθούν μέσα στα 10-15 χρόνια, πρέπει να το κάνουμε αυτό. Για τις ψηφιακές τεχνολογίες, εδώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο γιατί βλέπουμε ότι είναι πολύ γρήγορη η ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών και κυρίως πιστεύω θα υπάρξει και μεγαλύτερη σύνδεση με τις τεχνολογίες του διαστήματος σχετικά. Η Κάρη Μαντέλη έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πριν θέσω την ερώτησή μου θα ήθελα να εκφράσω την απογοήτευσή μου για τη σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εννέα μόνο γυναίκες εμείς ε, είχαμε κάνει τεράστιους αγώνες, αλλά εσείς ε, δεν φταίτε κύριε Σεύκοβιτς, οπότε εξ ονόματος των Πρασίνων σας, ε, σας καλωσορίζω. Και συνεχίζω στα γαλλικά, μιας και μιλάτε πολύ καλά. Η συμφωνία θα πρέπει να κλείσει, η συμφωνία 21, δηλαδή πάρα πολύ σύντομα. Έχουμε και τη συνάντηση κορυφής για το κλίμα ε, παρόλα αυτά το θέμα των μεταφορών δεν είναι κάτι το οποίο φαίνεται ιδιαίτερα στα πλαίσια της πολιτικής για το κλίμα, ενώ είναι κατεπήγοντα τα προβλήματα τα περιβαλλοντικά. Ε, έχετε ένα ξεκάθαρο οδικό χάρτη για τη συνάντηση αυτή κορυφής για το κλίμα. Η Επιτροπή είπε ότι υπάρχουν κάποια προγράμματα τα οποία εμείς θεωρούμε άχρηστα όπως η σύνδεση Λιών-Τωρίνο ε, είναι κάτι το οποίο έχει, θα αυξήσει το κόστος ε, άλλωστε και για τις μεταφορές πάρα πολύ ε, υψηλά. Έτσι κι αλλιώς έχουν υποεκτιμηθεί οι δαπάνες που θα απαιτηθούν κατά 30% τουλάχιστον, ενώ υπάρχουν πολλά να γίνουν για την βελτίωση της σύνδεσης ανάμεσα στις διαφορετικές περιοχές. Στη Γαλλία 8 εκατομμύρια Γάλλοι σαν παράδειγμα δεν έχουν πρόσβαση στις μεταφορές. Ε, βλέπετε λοιπόν ποιο είναι το πρόβλημα. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς χαρακτηρίζει και άλλες περιοχές της Ευρώπης. Και γιατί το Συμβούλιο και η Επιτροπή αυτά τα λίγα χρήματα θα τα χρησιμοποιήσουν για άχρηστους λόγους. Πώς μπορεί λοιπόν να χρηματοδοτεί αυτά τα άχρηστα προγράμματα όπως το Λιόν το Ρήνο ενώ θα μπορούσε και στα πλαίσια του RTE να δαπανίσει καλύτερα τα χρήματα, χωρίς όμως να γνωρίζουμε στην παρούσα φάση την οικονομική βιωσιμότητα του προγράμματος αυτού, όπως επίσης και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Πώς μπορεί λοιπόν από τη μία να σεβαστεί αυτό το 3% του ΑΕΠ που προβλέπεται από τις συνθήκες και από την άλλη ε, ε, τα προβλήματα, τα δημοσιονομικά που δημιουργούν τα σχέδια αυτά σε πολλές χώρες. Σας ευχαριστώ κυρία Ντέλη και για τα καλά σας λόγια στην αρχή της παρουσίασής σας. Αν μου επιτρέψετε τώρα θα συνεχίσω στα αγγλικά γιατί η ορολογία μου ε, σε σχέση με αυτούς τους νέους τομείς ε, είναι περιορισμένοι, αλλά συνεργαζόμενοι θα βελτιωθούν και οι γλωσσικές μου γνώσεις για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι η συνάντηση κορυφή στο Παρίσι για το κλίμα θα είναι ε, κρίσιμη. Ε, νομίζω ότι ακόμα και αν η Ευρώπη μπορεί πράγματι να κάνει περισσότερα από ό,τι έχει πετύχει μέχρι τώρα, ε, πάντα κάνουμε περισσότερα από τους άλλους ε, παγκόσμιους εταίρους μας, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάποια επιπλέον επιχειρήματα για να τους πείσουμε να πάρουν μέρος σε αυτήν την τεράστια προσπάθεια την οποία κάνουμε για να φροντίσουμε το κλίμα στον πλανήτη. Ο συνάδελφος Πότοτσεκ λέει ότι ο πλανήτης θα επιβιώσει των ανθρώπινων ενεργειών. Εμείς όμως θα επιβιώσουμε πάνω στον πλανήτη. Εδώ λοιπόν θα συμφωνήσω μαζί σας ότι απαιτείται να δείξουμε ότι είμαστε φιλόδοξοι και να πρέπει να έχουμε μια σφαιρική θα έλεγα αντιμετώπιση των προβλημάτων. Ενθαρρύνθηκα όταν είδα πάρα πολλές προσωπικότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις τελευταίες μέρες να δηλώνουν την αφοσίωσή τους προς τους στόχους αυτούς και νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα επηρεάσει τη συμμετοχή μας θετικά στο Παρίσι. Τώρα σχετικά με τα θέματα τα περιβαλλοντικά γενικότερα. Βλέπετε εδώ όλους τους στόχους τους οποίους έχουμε για το περιβάλλον. Ε, ε, στρατηγική 2020, στόχοι 2020, στόχοι 2030. Ξέρω ότι θα είμαστε επιτυχείς σε πολλούς τομείς, ε, λιγότερο ή περισσότερο. Νομίζω ότι και στις μεταφορές μέσω κάποιων κανονισμών, μέσω της πίεσης της βιομηχανίας να είναι πιο αποδοτική ενεργειακά, να χρησιμοποιήσει νέους τύπους ε, κινητήρες, Νομίζω ότι όλα αυτά έχουν βελτιώσει κάπως την κατάσταση. Οι στόχοι λοιπόν που έχουμε εδώ είναι δεσμευτικοί στόχοι όπως είπαμε, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει ε, να συνεχίσουμε τις πιέσεις έτσι ώστε να μειωθεί η μόλυνση. Δεν έχω χρόνο για τις υπόλοιπες ερωτήσεις, λυπάμαι. Λούγκρεν. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και ευχαριστώ κύριε Σεφκοβίτς που ήρθατε να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Θα ήθελα καταρχάς να κάνω κάποιες ε, ε, σκέψεις, να εκφράσω κάποιες σκέψεις για το βιογραφικό σας σημείωμα, το οποίο είναι εντυπωσιακό εν πολλής Αλλά από την άλλη με τρομάζει κιόλα. Από τότε που ήσασταν 18 δεν βλέπω να κάνετε ούτε μιας μέρας χειρονακτική δουλειά. Τώρα έρχεται να, κάνετε, να αναλάβετε καθήκοντα σε μια πολύ ψηλή θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου οι αποφάσεις θα επηρεάζουν την ε, ζωή και τη δουλειά εκατομμυρίων πολιτών, που εργάζονται στις μεταφορές, χωρίς να έχετε την παραμικρή εμπειρία από το χώρο αυτόν. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να πω ότι εγώ σου Σουηδός δεν θα μπορέσω να, σου, να εξηγήσω στους, ε, στο εκλογικό σώμα, κυρίως όσους ψηφοφόρους προέρχονται από τις μεταφορές, ότι ήσασταν ο καλύτερος ψήφισε τον τομέα αυτόν, γιατί δεν έχετε την παραμικρή εμπειρία. Και δεν γνωρίζετε τα σοβαρά προβλήματα του τομέα μεγαλώσατε και ανδρωθήκατε μέσα σε ένα χώρο με υψηλές σπουδέ, με πολιτική δραστηριότητα, με απίστευτους μισθού, μισθούς σε σχέση με αυτούς που υποτίθεται ότι θα εκπροσωπήσετε. Αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν να τα βγάλουν πέρα στο τέλος του μήνα ε, δεν καταλαβαίνω πώς θα τους εκπροσωπήσετε λοιπόν. Και κύριε Σεύκοβιτς, το πρόβλημα του κοινωνικού ντάμπινγκ είναι τεράστιο στον τομέα των μεταφορών. Ένα πρόβλημα το οποίο απορριθμίζει και αποδιαρθρώνει κάθε είδους ε, εταιρεία. Εμείς στην πατρίδα μου έχουμε για τις οδικές μεταφορές το πρόβλημα αλλοδαπών οδηγών φορτηγών, κυρίως από την Ανατολική Ευρώπη, οι οποίοι αναλαμβάνουν να κάνουν τις μεταφορές με τίμημα ε, τίμημα με το 1 τρίτο των δικών μας οδηγών. Κατοντάδες επιχειρήσεις μεταφορών έκλεισαν πέρυσι λόγω ακριβώς της απουσίας προστασίας εναντί αυτού του αθέμητου ανταγωνισμού στη Σουηδία. Οι επιχειρήσει μα δεν φοβούνται τον ανταγωνισμό, αλλά πρέπει αυτό να γίνεται σε όρου ισοδύναμου. Πώ μπορείτε λοιπόν να εξασφαλίσετε τέτοιου είδου ισότιμου όρου όταν το κοινωνικό ντάμπινγκ είναι ένας, ένα, ένα είδο πλεονεκτήματο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση και για τα ευγενή σας λόγια για το βιογραφικό μου σημείωμα. Σας βεβαιώνω όμως ότι γνωρίζω πολύ καλά τι σημαίνει χειρονακτική εργασία γιατί όταν ε, μεγάλωνα ως νέος είχα όπως κάθε νέος την ευκαιρία να εργάζομαι υποχρεωτικά τα καλά τους καλοκαιρινούς μήνες. Κάθε φοιτητή ήταν υποχρεωτικό να δουλεύει στα εργοστάσια. Το ίδιο συνέβη και όταν ήμουν μετά στη Ρωσία ως φοιτητή. Αυτό είναι μια εμπειρία που πολύ ευχαρίστω να μοιραστώ μαζί σας. Γνωρίζω λοιπόν πόσο σκληρή είναι αυτή η δουλειά και γνωρίζω με τι είδους στρες και άγχος δουλεύουν οι άνθρωποι αυτοί σε τέτοιες δύσκολες συνθήκες. Ιδιαίτερα δε στις οδικές μεταφορές, το κοινωνικό ντάμπινγκ είναι ασφαλώς ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Να αντιμετωπίσουμε. Αυτό που ήθελα λοιπόν ε, να σημειώσω, όπως είπα και στις αρχικές μου παρεμβάσεις, αλλά με χαρά θα το τονίσω και πάλι, είναι ότι θέλω μαζί με εσά να κοιτάξουμε εις βάθος και συνολικά το τι μπορεί να απλουστευθεί, το τι μπορεί να διευκρινιστεί ως προς τους κανόνες που εφαρμόζονται στις μεταφορές, γιατί όσο πιο απλοί είναι οι κανόνες, όσο πιο ξεκάθαροι, τόσο πιο ευχερής και η ε, ε, επιβολή τους και φαντάζομαι ότι θα μας στηρίξουν και οι κυβερνήσεις και οι αρχές που καλούνται να τηρήσουν και να εφαρμόσουν κανόνες αυτούς, έτσι ώστε να έχουμε απλούς κανόνες, σαφείς κανόνες, δίκαιους, ισοδίκαιους κανόνες και βέβαια από εκεί πέρα θα πρέπει οι εθνικές αρχές να μεριμνήσουν για την επιβολή τους. Τώρα για το πρόβλημα συγκεκριμένα των οδικών μεταφορών που αναφέρατε, εγώ πάλι μαζί με εσά. Θα είμαι διατεθειμένο να προτείνω στου κοινωνικού εταίρου την βελτίωση του κοινωνικού διαλόγου και την αναζήτηση μια λύση, η οποία παραδείγματι θα σήμαινε ε, το να μην χρειάζεται πάντοτε η παρέμβαση ε, στα θέματα των κοινωνικών δικαιωμάτων στις σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών στον χώρο των οδικών μεταφορών. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ απλό αυτό ώστε να μπορούμε να έχουμε μια ε, εφόσον βέβαια οι κανόνες είναι σαφείς και ευχερείς στην εφαρμογή τους για να έχουμε ένα σαφή και ε, σταθερό χώρο. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Τώρα περνάμε στο δεύτερο γύρο. Τρία λεπτά ερώτηση και απάντηση πάντα και οι κατευθύνες γραμμές είναι μία, ένα λεπτό για την ερώτηση και δύο λεπτά για την απάντηση. Παρακαλώ τηρήστε τον κανόνα αυτόν. Όσο πιο σαφή είστε και σύντομοι τόσο πιο διεξοδικά μπορεί να απαντήσει ο υποψήφιος επίτροπος. Ο κύριος Κόχ είναι τώρα επόμενο. Είναι πίσω σα κύριε Σέρκοβιτς, μην ψάχνετε στην αίθουσα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σεύκοβιτς, κάθομαι πίσω σας και ελπίζω μετά την ακρόαση να μπορώ να σταθώ στο πλευρό σας και να σας στηρίξω κι εγώ με την, με την ψήφο μου. Έχουμε λοιπόν ε, να μιλήσουμε για θέματα που έχουν να κάνουν με τις μεταφορές και με πάρα πολλά προβλήματα. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εκδώσει τη Λευκή Βίβλο με προγράμματα για τις μεταφορές, τις οδικές μεταφορές ε, και εδώ το θέμα μας είναι η ασφάλεια βέβαια και χιλιάδες νεκρών στους δρόμους ε, της Ευρώπης ε, ο στόχος λοιπόν της Λευκής Βίβλου ήταν να περιοριστούν ε, οι θάνατοι από τροχαία δυστυχήματα. Εγώ ήμουν εισηγητής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν ήρθε το θέμα στην έκθεση και θα ήθελα να σας ρωτήσω τι είδους συγκεκριμένα μέτρα σκοπεύετε να λάβετε εφόσον επιβεβαιωθείτε στη θέση του Επιτρόπου προκειμένου να εκμηδενίσετε τον κίνδυνο των τροχαίων δυστυχημάτων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κόχ για την ερώτησή σας. Έχει τεράστια σημασία πιστεύω για εκατοντάδες χιλιάδων Ευρωπαίους όχι μόνο 26.000 νεκροί πέρσι, 250.000 σοβαρά τραυματίες επίσης καταγράφηκαν σε ε, τροχέα το 2013 και μπορεί να λέμε ότι είναι η πιο ασφαλής, ο πιο ασφαλής χώρος των μεταφορών η Ευρώπη, αλλά σε απόλυτους όρους τα στοιχεία αυτά είναι απαράδεκτα υψηλά. Αλλά να δούμε λίγο τα στοιχεία. Το 2014 παρότι είχαμε πολύ σταθερή μειωτική τάση, ως προς τον αριθμό των θυμάτων των τροχαίων τα τελευταία χρόνια με μείωση κατά 18% βλέπουμε ότι το 2014 μπορεί να εμφανιστεί μια ελαφρά αύξηση των στατιστικών στοιχείων. Θα πρέπει να δούμε γιατί συνέβη αυτό. Υπάρχουν λόγοι όπως οι παραδείγματι πολύ ε, μακρύς ή άλλοι παράγοντες. Ε, πάντως είναι ανησυχητικά τα στοιχεία. Και ήδη αυτό που ε, έχει φέρει καρπούς είναι η αναζήτηση των λόγων και βέβαια πρέπει από εδώ και πέρα να κοιτάξουμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Αφενός μεν θα πρέπει να εφαρμοστεί η οδηγία ε, η σχετική με την ασφάλεια στις οδικές μεταφορές, ε, επί παραδείγματι οδηγοί οι οποίοι μέχρι τώρα οδηγούσαν ε, κατά τρόπο επικίνδυνο επειδή βρίσκονταν έξω από τα σύνορα τα οδικά της χώρας τους, τώρα θα κινδυνεύουν με πρόστιμο και εφόσον έχουν παραβιάσει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας σε ξένες χώρες. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα. Μπορούμε επίσης να δούμε άλλους τρόπους να μειώσουμε τα σοβαρά, τους σοβαρούς τραυματισμούς που προκύπτουν από τα τροχέα ε, και πολλά άλλα θετικά μέτρα που μπορούμε να αναλάβουμε στα αστικά κέντρα με νέες ε, προσεγγίσεις και λύσεις οι οποίες θα μπορούσαν να διευκολύνουν ε, ακόμη και αυτόν που έχει εμπλεκεί, αυτόν έχει εμπλεκεί κάποιο σε ένα ατύχημα, να βοηθήσουν στην ταχεία αντιμετώπιση των προβλημάτων. Ο κύριος Σασόλη έχει το λόγο, χωρίς μικρόφωνο. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ζητήσω από τον υποψήφιο Επίτροπο να του θυμίσω μάλλον ότι στην τελευταία συνάντηση που πήραν μέρος οι συντονιστές της Επιτροπής Μεταφορών και οι εισηγητές για το τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο ε, συζητήθηκε να δοθεί στο Κοινοβούλιο ε, η εντολή διαπραγμάτευσης ε, και του τεχνικού πυλώνα αλλά και του πολιτικού πυλώνα. Πιστεύετε κύριε Επίτροπε ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Πιστεύετε ότι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον προηγούμενο Φεβρουάριο μπορεί να αντιπροσωπεύσει την σωστή διαπραγματευτική βάση για τους επερχόμενους τριμερείς διαλόγους. Δεύτερη ερώτηση. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει να υιοθετήσει το 2015 την αλλαγή του κανονισμού ΕΑΣΑ, εάν σε αυτή την περίπτωση είναι καταφατική η, απόφαση, η απάντησή σας, Πώς θα ξεκινήσετε ε, τις διαπραγματεύσεις αυτές για το ΣΥΝ 2. Σας ευχαριστώ και εύχομαι καλή δουλειά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σασόλη για τις ερωτήσεις σας. Είναι θέματα τα οποία πράγματι βρίσκονται στο τραπέζι το νομοθετικό στην παρούσα φάση και είναι ένα θέμα στο οποίο καλούμε εφόσον πρόταθω να ασχοληθώ γρήγορα. Η Ιταλική Προεδρία υποστηρίζει ιδιαίτερα το πακέτο το σειροδρομικό. Έχουν προσφέρει πάρα πολλά στην διαπραγμάτευση. Έχουν υπάρξει, ε, προβλέπεται να υπάρξει συνάντηση των αρμόδιων Υπουργών Μεταφορών για το θέμα αυτό και οι Υπουργοί θα πρέπει ε, να στηρίξουν την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την σοφή κατεμέ τη συνοχή αυτών των προτάσεων σε ένα πακέτο. Έχουν υπάρξει βήματα προόδου σε επίπεδο τεχνικό. Βέβαια υπάρχουν τεχνικά προβλήματα τα οποία λειτουργούν ως τροχοπέδι για την σειροδρομική βιομηχανία. Αλλά θα πρέπει και στο πολιτικό κομμάτι να κάνουμε βήματα προόδου η ανάπτυξη μέσων εμπιστοσύνης, δημιουργίας εμπιστοσύνης, κλίματος εμπιστοσύνης νομίζω ότι θα μας οδηγήσει σε σωστές λύσεις οι οποίες θα είναι αποδεκτές από την πλειοψηφία της Επιτροπής σας και του συνόλου της Ολομέλειάς σας. Είμαι βέβαιος ότι θα προχωρήσουμε και με την αναθεώρηση του ΕΑΣΑ ε, όχι ότι δεν κάνει πολύ καλή δουλειά η ΕΑΣΑ, υπάρχουν εξαιρετικά άτομα εκεί που κρατούν την ασφάλεια στις πτήσεις στο ίδιο επίπεδο με τη ΣΥΠΑ. Θα θέλαμε όμως να, να αντιμετωπίσουμε τις μελλοντικές προκλήσεις και η πρόοδος στο πακέτο ΣΥΝ2 θα δώσει δυνατότητες περαιτέρω βελτίωσης. Μαρινέσκου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, αναφερθήκατε ήδη στον, στους ενίους εθέρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εγχείρημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά φυσικά πρέπει και τα κράτη-μέλη να πιστούν να σταματήσουν την στεναρή αντίδραση που έχουν δείξει για να γίνει πραγματικότητα αυτό το εγχείρημα των ενιαίων εθέρων. Πρέπει για να γίνει αυτό πραγματικότητα να εφαρμοστεί το ΣΕΣΑΡ. Το ερώτημα είναι πώς θεωρείτε ότι θα μπορέσετε να εξασφαλίσετε την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών και του σχεδίου ΣΕΣΑΡ και πάλι είναι ένα ευρωπαϊκό εγχείρημα ώστε να μπορέσουμε με τον τρόπο αυτό να επιτύχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στον εναέριο έλεγχο πάνω από την Ευρώπη. Ένα ακόμα <clears throat> ερώτημα για το πρόγραμμα έγνος καλύπτει το σύνολο του ευρωπαϊκού χώρου ως διαστημικό πρόγραμμα, τότε θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ τις ε, διαδικασίες προσγείωσης στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Πότε νομίζετε ότι θα μπορέσει να χρησιμοποιεί το πρόγραμμα έγνωση από τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια και επίσης για, το, για τις κοινωνικές συνθήκες τι άποψη έχετε για τα πρόστιμα που χρειάστηκε να πληρώσουν οι οδηγοί φορτηγών που έχουν ξεπεράσει το χρόνο που περνάνε μάλλον το χρόνο ανάπαυσής τους στις καμπίνες των φορτηγών, χάρη αυτό στη Γαλλία. Και αν θέλετε μπορώ να, να σας πω πώς ήταν τα πράγματα και στη δική μου χώρα πριν πέσει το σιδηρούν παραπέτασμα. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Μαρινέσκου. Πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικό γιατί είσαστε πραγματικά εμπειρογνώμων, υπήρξατε υπουργό μεταφορών και είστε και μηχανολόγος. Το πρώτο ερώτημά μου, η ερώτημά σας, συγγνώμη. Δεν μπορώ να μην πω ότι νιώθω μεγάλη ματέωση για το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει πρόοδος για τα λεγόμενα block εθέρων. Είμαστε πολύ μακριά από το να έχουμε ένα σύστημα που θα μοιάζει με το σύστημα των ΗΠΑ που είναι ενιαίος ο ενάριος χώρος. Ελπίζω όμως ότι αυτά τα εννέα λειτουργικά τμήματα του εναερίου χώρου θα μπορέσουν να γίνουν, νόμιζα θα γίνουν πραγματικότητα, αλλά ούτε και αυτό έχει καταστεί δυνατό. Δεν υπάρχει λογική εξήγηση για μένα για αυτό το γεγονός. Αν θέλουμε να χάνουμε 5 ε, εκατομμύρια ευρώ το χρόνο επειδή δεν θέλουμε να βελτιώσουμε το σύστημα, είναι πραγματικά απώλεια χρημάτων. Το ΣΕΖΑ θα μπορούσε να βοηθήσει γιατί και εξάλλου έχει αξιολογηθεί πολύ θετικά από τους ανταγωνιστές μας. Ξέρουμε ότι κάποιες ασιατικές χώρες έχουν ενδιαφερθεί ιδιαίτερα για το σχέδιο ΣΕΖΑ. Είναι πιο <clears throat> αποτελεσματικό, επιτρέπει τα αεροπλάνα να πετούν πιο κοντά το ένα το άλλο, να υπάρχει καλύτερη χρησιμοποίηση του εναέριου χώρου και εξασφαλίζει και μεγαλύτερη ασφάλεια για τα αεροδρόμια. Για να κλείσω λοιπόν αυτό το σημείο, θα προχωρήσω στο διορισμό ενός μάνατζερ ανάπτυξης για το ΣΕΣΑΡ που ελπίζω ότι θα προωθήσει σε πραγματική εφαρμογή αυτό το σχέδιο στην Ευρώπη και συγγνώμη τελείωσε ο χρόνος μου. Ναι, φταίει η ερώτηση που ήταν πάρα πολύ μακροσκελής. Κύριε Ταπαρντέλ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, το δικό μου ερώτημα είναι πιο άμεσο και πιο συγκεκριμένο. Αφορά το τέταρτο σιδηροδρομικό σχέδιο σε ό,τι αφορά τον πολιτικό πυλόν αυτού του πακέτου. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψή σα σε σχέση με την πρόθεση του τομέα αυτού. <clears throat> Υποστηρίζετε την αρχή του, του ανταγωνισμού και για τον τουρισμό. Ξέρω ότι δεν είναι αυτό το τμήμα της αρμοδιότητάς σας, αλλά γνωρίζετε ότι υπάρχει στενή σχέση μεταξύ μεταφορών και τουρισμού. Υπάρχουν πολλές ελκυστικές περιοχές για τον τουρισμό στην Ευρώπη, αλλά δεν έχουν την απαραίτητη προσβασιμότητα όπως οι μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Γιατί, Γιατί δεν έχουν τις απαραίτητες υποδομές. Τι στρατηγική θεωρείτε ότι, να, ότι πρέπει να εφαρμοστεί για να υπάρξει μια μεγαλύτερη ανάπτυξη των υποδομών μεταφορών στις περιοχές αυτές που έχουν μεγάλο δυναμικό για τον τουρισμό, γιατί ξέρετε ότι ο τουρισμός παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του ΑΕΠ της ευρωπαϊκής οικονομίας και είναι απαραίτητε μεταφορέ για τον τουρισμό. Τρίτο ερώτημα. Τι θα γίνει με τα κράτη-μέλη που βρίσκονται στα ανατολικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω τη Ρουμανία, τη χώρα από την οποία προέρχομαι εγώ. Οι χώρε αυτέ είναι συνδεδεμένες με χώρες έξω από την Ευρώπη, με την Κίνα, τη Ρωσία, την Αποανατολή τι στρατηγικέ θα πρέπει να εφαρμοστεί στι χώρε αυτέ για να αναπτύξουν περαιτέρω στα σύνορά του τι υποδομέ του μεταφορών. Και με τον τρόπο αυτό θα μπορούμε να έχουμε καλύτερη σύνδεση με του ανατολικού μα ε, γείτονε, όχι μόνο σε επίπεδο μεταφορών, αλλά σε και επίπεδο οικονομικών σχέσεων. Οι μεταφορέ λοιπόν με τι υποδομέ και την ε, λειτουργία τη είναι ένα από του πυλώνε Ευρωπαϊκή Ένωση και κλείνοντα. Πρέπει να πω ότι είναι λίγε οι γυναίκες που είναι ε, <clears throat> επίτροποι, αλλά έχουμε πολλές γυναίκε στην Επιτροπή Μεταφορών και αυτό είναι θετικό. Μένει ένα λεπτό μονάχα για τον ε, Επίτροπο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, εάν δεν λάβετε όλες τις απαντήσεις που περιμένετε θα είναι δική ευθύνη διότι δεν ε, αφήσατε αρκετό χρόνο, μιλήσατε πάρα πολύ ώρα. Όπως είχα πει, ούκεν το πολλό το εφ και ως εκ τούτου θα δώσω στον Επίτροπο το λόγο για όσο χρόνο περισσεύει τώρα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα χρειαστεί μια ιδιαίτερη διμερή συνάντηση για όλες αυτές τις ερωτήσεις από ό,τι διαπιστώνω. Πάντως θα ήθελα να πω ότι για το πακέτο για τους σιδηροδρόμους θα πρέπει να βρούμε μια λύση αποδεκτή για την πλειονότητα των ε, κρατών μελών και βέβαια την πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, με λύσεις ε, διαφορετικές και ποικίλε τις οποίες είναι τεθειμένος να εξετάσω στο σύνολό τους, αλλά υπάρχουν πολλά έχει σημασία να εξασφαλιστεί πρόοδος. Θα πρέπει επίση να αναπτύξουμε τι δυνατότητε που μα δίνουν τα ερθωτικά ταμεία και εδώ έχουν ευθύνη τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να δούμε πόσο ποιοτικέ ε, υποδομέ μεταφορών μπορούμε να έχουμε στην Ευρώπη, γιατί γνωρίζει κανεί ότι θα ταξιδέψει κάπου με τρόπο ασφαλή και ευχερή και μπορούμε χάρη στα ερωτικά ταμεία να προωθήσουμε και τα τουριστικά αξιοθέατα στις ε, χώρες μας. Αυτό θα είναι πολύ σοβαρή επένδυση για το μέλλον, ο Πρόεδρος. Τέρμα, θα πρέπει δυστυχώς για να είμαι δίκαιος προς όλους να σας διακόψω. Δεν είναι δική σας ευθύνη βέβαια. Α, ο κύριος Κλούν έχει το λόγο. Κυρία Κλούν. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα ίσως να βοηθήσω με τις ε, ερωτήσεις της συνάδελφο για να πάρουμε τις απαντήσεις. Ε, θα θέλαμε σε σχέση με τις απομονωμένες και τις πιο απομακρυσμένες ε, περιοχές της ε, περιφέρειας ή το υπαίθρου της Ευρώπης να μιλήσουμε όταν υπάρχουν εκεί αεροδρόμια τα οποία μπορούν να βοηθήσουν βέβαια και για την πρόσβαση σε τουριστικά αξιοθέματα κτλ. Θα πρέπει να βοηθήσουμε λοιπόν στα περιφερειακά αεροδρόμια που κινδυνεύουν με κλείσιμο να διαφυλαχθούν. Οι κρατικές ενισχύσεις και οι σχετικοί κανόνες πρέπει να αξιολογηθούν βεβαίως, αλλά δεν θέλω να μου πείτε ποιες είναι οι προτεραιότητες σε σχέση με τα περιφερειακά αεροδρόμια και τα προβλήματα, όπως αναφέρω, των περιφερειακών, των απομονωμένων και των ισοτικών περιοχών της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι τοπικές περιφερειακές αεροπορικές συνδέσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένως και τα περιφερειακά αεροδρόμια αλλά θα πρέπει να δούμε ποια είναι η ικανότητα, η χωρητικότητα των αεροδρομίων αυτών στην Ευρώπη και άμα δείτε και τη γειτονιά μας βλέπετε ότι η γειτονιά μας προχωράει με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Αν δείτε το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης που σύντομα θα μπορεί να υποδέχεται 140-150 εκατομμύρια επιβάτες το χρόνο. Μα βλέπετε τι γίνεται στο Ντουμπάι όπου αυτός ο αριθμός μπορεί να φτάσει στα 160 εκατομμύρια επιβάτες τον ε, χρόνο, ενώ στο Χήθρο έχουμε μονάχα 70 εκατομμύρια το maximum, <clears throat> βλέπετε ότι οι εξελίξεις στην ε, Μέση Ανατολή και στη γειτονιά μας είναι τόσο έντονες που θα πρέπει να τις λάβουμε υπόψη μας και θα πρέπει να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα αεροδρόμια μας και πώς αντιμετωπίζουμε τις αεναερίες μεταφορές ως σύνολο. Φυσικά είναι σημαντική η αύξηση της αποδοτικότητας στον αέρα και στα αεροδρόμια. Πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε μια καλή λύση για να αναπτύξουμε το πακέτο για την χωρητικότητα των αεροδρομίων. Πιστεύουμε ότι αν, εφαρμόσουμε τις, αν εφαρμοστούν οι προτάσεις που έχουμε κάνει και ξέρω βέβαια και ποια είναι τα προβλήματα που εμπεριέχουν, μπορούμε να αυξήσουμε τη χωρητικότητα των αεροπολικών των αεροδρομίων στην Ευρώπη κατά 20 εκατομμύρια επιβάσεις το χρόνο χωρίς να προσθέσουμε ούτε ένα διάδρομο απογείωσης προσγείωσης. Πρέπει λοιπόν να εγκριθεί αυτό το πακέτο σε σχέση με τις κρατικές επιδοτήσεις, νομίζω ότι οι κατευθυντέριες γραμμές για τις επιδοτήσεις που εγκρίθηκαν πρόσφατα είναι πολύ θετικές. Είναι καλό που ότι τις έχουμε. Γιατί ξέρω ότι αργότερα θα συζητήσετε και την κατάσταση των λιμένων και πιστεύω ότι σε ό,τι αφορά τα αεροδρόμια τουλάχιστον έχουμε καλούς κανόνες για να αξιολογούμε τις κρατικές επιδοτήσεις και αυτό θα είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία θέλω να συζητήσω μαζί με την κυρία Βέσταγκερ, την συνάδελφό μου που θα είναι αρμόδια για τις, ελπίζω για τα θέματα ανταγωνισμού και που θα καλύπτει και τις μεταφορές. Ο κύριος Πορέμπα έχει τώρα το λόγο, ο είναι και αυτός πίσω σας. Κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα δύο πράγματα να σας ρωτήσω κύριε Επίτροπε σχετικά με το δίκτυα στην Ανατολική Ευρώπη. Καταρχάς, ο δικός άξον Βία Καρπάτια που ε, εκινεί στην Λιθουανία και περνά από την Σλοβακία, την Τσεχία και καταλήγει στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς δεν συμπεριλήφθη στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Αλλά υπάρχει μια πολιτική πρωτοβουλία εδώ από τις περιφέρειες αυτές έτσι ώστε να χρηματοδοτηθεί και στα πλαίσια του Connecting Europe αν είναι δυνατόν. Πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί. Θα βοηθήσετε έτσι ώστε να δοθεί στο μέλλον μια επιτυχής κατάληξη σε αυτή την προσπάθεια γιατί αυτός ο οδικός άξον είναι από τους πιο σημαντικούς παράγοντες ανάπτυξης της περιοχής. Τώρα, συνοπτικά οι σιδηρόδρομοι ε, τους οποίους ε, θα χαράξει η Ρωσική Ομοσπονδία μέσω Σλοβακίας και Αυστρίας. European funds. Thank you. Thank very much, Mr. for... <coughs> Ευχαριστώ κύριε Πορέμπα και για τις δύο ερωτήσεις σας. Σχετικά με την Βία Καρπάτια, είναι αλήθεια ότι δεν έχει συμπεριληφθεί στα TENS αλλά έχει συμπεριληφθεί στο λεγόμενο συνολικό δίκτυο, ολοκληρωμένο καλύτερα δίκτυο το, και αυτό δείχνει την σημασία που έχει η ανάπτυξη των, των μεταφορών στην Ευρώπη σε αυτή την περιοχή ιδιαίτερα. Θα πρέπει λοιπόν να συνδυάσουμε ε, και τα ταμεία συνοχής τα οποία έχουν στην δυνατότητά τους οι χώρες αυτές γνωρίζετε ότι υπάρχει ένα κριτήριο που λέει ότι αν σε αυτό το συνολικό δίκτυο υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί σαν ε, ε, ευρύτερης ευρωπαϊκής σημασίας και διαμεθοριακά μεγάλης σημασίας. Νομίζω λοιπόν ότι στην περίπτωση αυτή μπορούμε να βρούμε μια λύση. Αυτό το οποίο πρέπει να επιδιώξουμε στην Ανατολική Ευρώπη είναι η ποιότητα του προγράμματος ή η δυνατότητα απορρόφησης των πιστώσεων που είναι διαθέσιμα για τα διαφορετικά ταμεία στις χώρες αυτές και η ταχύτητα γενικά σχεδίασης. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι αν δεν υπάρξει αυτή η προσπάθεια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι πιστώσεις του Ταμείου Συνοχής. Μιλήσατε για τα δικαιώματα των επιβατών σε όλους τους τομείς των μεταφορών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμένει σε αυτά και είχαμε και μια συμφωνία διακομματική γύρω από αυτό. Ποια είναι η άποψή σας για το ψήφισμα του Κοινοβουλίου του 2012 και του 2011 για τα δικαιώματα των επιβατών και αυτών με μειωμένη κινητικότητα που θα πρέπει να ενημερώνονται σωστά σε σχέση ε, και με ε, τα δρομολόγια και στις αερομεταφορές ε, και θα πρέπει να μην υπάρχουν εξαιρέσεις από την ευθύνη των αερομεταφορέων στην περίπτωση καθυστερήσεων για τεχνικούς ή άλλους λόγους. Σαν παράδειγμα θα το πω ότι έχουμε κάνει κάποια βήματα στον τομέα των δικαιωμάτων αλλά δυστυχώς πολλά μένει να γίνουν και το ίδιο θα πρέπει να ισχύσει επίσης και για τα νυχτερινά τρένα. Uh, τα δικαιώματα των επιβατών έχετε ε, πολύ σωστά που αναφέρεστε στον όρο «We've come a long way», διανύσαμε ένα μεγάλο κομμάτι του δρόμου. Πράγματι έχετε πιέσει σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε τα δικαιώματα των ταξιδιωτών να είναι σε ε, εξέχουσα θέση. Το επόμενο βήμα τώρα. Το επόμενο βήμα είναι να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε πόσο τα δικαιώματα των επιβατών θα ενταχθούν στα πλαίσια των νέων διατροπικών μορφών μεταφορών αν αλλάζει κανείς σαν παράδειγμα μέσο από τρένο σε αεροπλάνο ή σε πλοίο κτλ θα πρέπει να διατηρείται ο σεβασμός των δικαιωμάτων. Αυτό το οποίο με απασχολεί ε, βλέπουμε ότι μόνο το 5% των επιβατών αυτή τη στιγμή έχουν αποζημιωθεί σαν παράδειγμα στην περίπτωση που έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά τους. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε ένα σωστό μηχανισμό επιβολής και γιατί είναι περίπλοκοι οι κανόνες αλλά και γιατί όπως σας είπα δεν έχουμε την δυνατότητα να επιβάλλουμε το σεβασμό των κανόνων αυτών στα κράτη-μέλη. Πρέπει λοιπόν σιγά σιγά να αντιμετωπίσουμε τις παραβάσεις αυτές, τις καθυστερήσεις αυτές, έτσι ώστε οι πολίτες να ξέρουν πού πρέπει να προσφύγουν και να μην εξαρτώνται μόνο από την τοπική δικαιοσύνη για να αποζημιωθούν για την παραβίαση των δικαιωμάτων τους για τους επιβάτες μειωμένης κινητικότητας. Εδώ θα συνεργαστώ με την κυρία Τίσεν ε, για την Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας που θα δίδει με το νόμο την εγγύηση ότι οι επιβάτες αυτοί θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλους τους άλλους ε, επιβάτες. Και θα ήθελα να αναφερθώ και στις πληροφορίες που μπορεί να πάρει κανείς από το διαδίκτυο, από την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές ακόμα και αυτοί που έχουν προβλήματα όρασης μέσω των smartphones, των εφιών κινητών τηλεφώνων. Η κυρία Τσέσκουν Μπιλμπάου Μπαραντίκα Ευχαριστώ κύριε Σεύκοβιτς. Το τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι δεν ευδοκίμησε το τρίτο. Το να υπάρχει μια νέα διακυβέρνηση στις μεταφορές που ξεπερνάει τα ιστορικά μονοπόλια και τις εθνικά στεγανά, θέλετε να το κάνετε αυτό. Υπάρχει μια συμφωνία στο Κοινοβούλιο για τις έξι εκθέσεις, αλλά το Συμβούλιο δεν έχει καταλήξει σε συμφωνία θίγει τι εταιρείε που θέλουν ασφάλεια δικαίου και αυξάνει το κόστο τη γραφειοκρατίας. Αν αυτή η κατάσταση συνεχίσει να λειτουργεί έτσι, ε, είσαστε έτοιμοι να προχωρήσετε στην οδηγία, στην εφαρμογή τη οδηγία για τη διαλειτουργικότητα χωρί πολιτική υποστήριξη. Θα κάνετε μελέτε για να δείτε ποιε είναι οι συνέπειε που θα αποκύψουν από το τέταρτο πακέτο για τι επενδύσει και την απασχόληση. Τι θα γίνει αν δεν εγκριθεί για αυτά που ανέφερα και για την καινοτομία και την διαλειτουργικότητα στο σιδηροδρόμο. Και τέταρτον, πώ θα υποστηρίξετε το shift to rail, αυτό το κοινό εγχείρημα που είναι σημαντικό για του σιδηροδρόμου. Και τέλο, τι πιστεύετε για την διαχείριση, το, για την διάκριση μεταξύ διαχειριστών υποδομών και των αυτών που λειτουργούν τι σιδηροδρομικέ γραμμέ. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριο Σεύκοβιτ. Σας ευχαριστώ για τα ερωτήματά σα γιατί νομίζω ότι βρίσκονται στον πυρήνα των διαπραγματεύσεων για το τέταρτο συνδρομικό πακέτο. Αν ήξερα όλες τις απαντήσεις για αυτά θα ήμασταν πολύ κοντά. Αλλά μπορώ να σας δώσω τη δική μου αίσθηση όπως βλέπω τώρα τα πράγματα. Η πρώτη προτεραιότητα για μένα είναι να διατηρηθεί ω σύνολο αυτό το πακέτο. Γιατί νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε πολύ καλά στα, έχουμε προχωρήσει καλά στα τεχνικά στοιχεία του πακέτου, αλλά θα ήταν κρίμα λόγω τη πρόοδου στο τεχνικό επίπεδο και των προβλημάτων που έχουμε στο πολιτικό επίπεδο, το επίπεδο διακυβέρνηση, να εγκαταλείψουμε αυτό το πακέτο. Για να είμαι ειλικρινή, δεν θέλω να έρθω ενώπιον σα με ένα πέμπτο σιδηροδρομικό πακέτο. Θα είμαι πολύ ικανοποιημένο αν το τέταρτο πακέτο είναι το τελευταίο για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και αν μπορούμε να ξεπεράσουμε τα θέματα τα οποία ακόμα δεν έχουν επιληθεί. Μπορούμε να έχουμε διαφορετικά υποδείγματα. Έχουμε υποδείγματα που υπάρχει πλήρης ε, ε, διάκριση μεταξύ του παρόχου υπηρεσιών μεταφορών και του διαχειριστή των υποδομών, που έχει δώσει πολύ καλά αποτελέσματα. σε ορισμένα κράτη-μέλη αυτό είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται ως μια κίνηση που θα έθετε σε κίνδυνο την απασχόληση στον ε, <clears throat> σιδηροδρομικό χώρο και την και δυσκολίε για τι εταιρείε αυτέ. Είμαι έτοιμο να ακούσω αυτέ τι προτάσει. Αυτό που με ενδιαφέρει όμω είναι η ισότητα ανταγωνισμού, η δημοσιονομική διαφάνεια και η κοινή κατανόηση ότι αυτό είναι ο τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Προφανώ θα πρέπει να υπάρξει και μια μεταβατική περίοδο που θα εξασφαλίσει την ισότητα ανταγωνισμού για όλου του συνδρομικού φορεί και με τον τρόπο αυτό μπορούμε να βάλουμε σε νέε ράγες τον συνδυοδομικό τομέα στην Ευρώπη και δεν θα χρειαστεί να προχωρήσουμε και σε πέμπτο συνδυοδομικό πακέτο. Ο Λούις Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε υποψήφοι ε, Επίτροπε ε, κανονικά θα πρέπει να μετατρέψουμε τις ιερομικές μεταφορές και να τις κάνουμε αποδοτικές ενεργειακά ε, και ε, εποφελείς για τις επιχειρήσεις και για τους ε, επιβάτες δεν έχουν το ποσοστό στις μεταφορές συνολικά το οποίο τους αξίζει. Υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια στη σωστή τους ανάπτυξη. Υπάρχει και αντίσταση από διάφορες χώρες που ε, εμένουν να κρατούν τις αρμοδιότητες τους γύρω από τη ρύθμιση των σιωδρομικών μεταφορών. Ε, με το άνοιγμα των εθνικών αγορών θα πρέπει να μην ε, παρεμποδίζουν ε, την είσοδο στην αγορά κάποιων εταιριών και δεν θα πρέπει να ενισχύουν τις παραδοσιακές ιοδρομικές εταιρείες που ελέγχουν και έχουν τα μονοπόλια. Και τι γίνεται με τις λεγόμενες ρήτρε αμοιβαιότητας στον τομέα των σειοδρομικών μεταφορών. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας, είναι πεθεμητή. Νομίζω ότι ε, μου δίδεται τα επιχειρήματα για να προωθήσω και τα δύο τμήματα του πακέτου από κοινού. Δηλαδή απαιτείται πρόοδο στο τεχνικό κομμάτι, απαιτείται όμως και πρόοδος στον τομέα τον τεχνικό. Τα κράτη-μέλη και οι εταιρείες δεν θα πρέπει να νιώθουν ότι δεν υπάρχει σωστός ανταγωνισμός και ότι υπάρχουν στρεβλώσεις εις βάρος τους σε κάποιες χώρες μπορεί να έχουν υπάρξει αναθέσεις ε, επιχειρηματικών σιωδρομικών δραστηριοτήτων χωρίς ε, δημόσιους διαγωνισμούς και διαδικασίες. Οπότε σε αυτή την περίπτωση και εφόσον δεν υπάρχει και η απαιτούμενη διαφάνεια δημιουργείται η αίσθηση ότι τα χρήματα τα οποία δίδονται στις επιχειρήσεις τις οδρομικές για τη διαχείριση των υποδομών χρησιμοποιούνται ουσιαστικά για την ενίσχυση της επιχειρηματικής τους θέσης. και χρησιμοποιούν τα χρήματα αυτά για την εξαγορά επιχειρήσεων ανταγωνιστικών σε όμορες χώρες. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, πρέπει να αντιμετωπιστεί και μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο μέσω της σωστής διαδικασίας διαφάνειας και ξεκάθαρων κανόνων. Έχω την ελπίδα ότι μετά από μια μεταβατική περίοδο η οποία δεν θα είναι ιδιαίτερος μακρά θα γίνουν οι ρυθμίσεις αυτές γιατί αλλιώς φοβάμαι ότι αν περάσουμε στην εφαρμογή των κανόνων γύρω από τις ρήτρε αμοιβαιότητας θα δημιουργήσουμε το αντίθετο αποτέλεσμα. Αντί να ολοκληρώσουμε δηλαδή την αγορά, αντί να δημιουργήσουμε μια πραγματικά ενιαία ευρωπαϊκή περιοχή σιδηροδρόμων, θα αρχίσουμε μια διαδικασία πολυδιάσπασης και δημιουργίας νέων εμποδίων και αυτό θα πρέπει να το αποφύγουμε με κάθε κόστος. Θα ήθελα να σας καλέσω λοιπόν όλους και ιδιαίτερα το Συμβούλιο να επιλέξει μια σωστή και δίκαιη λύση και για τα πολιτικά προβλήματα και για τα τεχνικά. Κυρία Γιάννα Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Σεύκοβιτς. Η επενδύση του κύριου Γιάνκερ έχουν σε στόχο ανάκαμψη και απασχόληση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει ένα προϋπολογισμό 30 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις ε, επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Πρέπει όμως να δαπανηθούν. Με, τις ε, κρίσεις, με την κρίση τα ευρωπαϊκά κράτη δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν αυτά τα σχέδια. Είσαστε έτοιμος να εξασφαλίσετε την απαραίτητη ευκαμψία ώστε αυτές οι επενδύσεις να μην καταλογίζονται στο, στο χρέος των κρατών μιλών και επίσης πώς θα αντιμετωπίσει τα κάτι μελη τα οποία εμποδίζουν τις διαμεθοριακές μεταφορές όπως γίνεται στη δική μου χώρα στα κεντρικά πυρηναία και για την απασχόληση. Είναι απαραίτητο να υπάρξει ένα κοινωνικό πακέτο για τους εργαζόμενους στον τομέα των μεταφορών. Έχουμε τους ναυτικούς, έχουμε τους οδηγούς φορτηγών και έχουμε κοινωνικό ντάμπινγκ το οποίο θίγει πια και τους πιλότους των αεροπορικών εταιριών. Πώς Πότε θα μπορούμε να περιμένουμε από εσά, κύριε Επίτροπε, να παρουσιάσετε ένα πακέτο για το κοινωνικό τάμπινγκ ενώπιον του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ και για τα δύο ερωτήματα. Το πακέτο επενδύσεων που αναφερθήκαμε προηγουμένω. είχα πει ότι είναι μια σαφή ε, δέσμευση του Προέδρου της Κομισιόν ότι πολύ σύντομα θα πρέπει να έρθουμε ενώπιόν σας μέσα σε τρεις μήνες για να σας προτείνουμε τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτό το πακέτο 300 δισεκατομμύριων για επενδύσεις. Και εδώ εγώ είμαι απλώς ένας υποψήφιος επίτροπος. Αν πράγματι αναλάβω το, τα θέματα μεταφορών και διαστήματος, είναι πολύ σαφές το κονδύλιο που θα πάει στις μεταφορές. Πιστεύω επίσης ότι σε αυτό το χώρο θα έχουμε σχέδια τα οποία θα είναι πολύ ελκυστικά για ιδιωτικούς επενδυτές σε εταιρική σχέση δημόσια, δημόσιου και ιδιωτικού χώρου και επίσης θα μπορέσουμε να τα συζητήσουμε αυτά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που μπορεί να πράξει περισσότερα στον τομέα αυτό αλλά επίσης και τα συνταξιοδοτικά ταμεία, οι ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν τα χρήματα μπορεί να προσελκυστούν και να επενδύσουν και αυτές για αυτά τα προγράμματα υποδομών. Τώρα, εάν πρόκειται για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει συζητηθεί πολλές φορές. Το Σύμφωνο Σταθερότητας έχει ήδη τροποποιηθεί και υπάρχουν ρήτρε ευκαμψίες που έχουν τροποποιήσει την αρχική μορφή αυτού του συμφώνου. Πιστεύω ότι θα πρέπει να βρούμε τους τρόπους με τους οποίους να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις επενδύσεις από τους δημόσιους πόρους και να εξακολουθήσουμε να έχουμε μία δυνατότητα χωρίς να θίξουμε το δημόσιο χρέος. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για την επερχόμενη Κομισιόν. Είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Μοσκοβιτσί και ο κύριος Κατάινα καθώς και ο κύριος Δομπρόφσκης θα αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό. Ελπίζω ότι ακόμα και στο τωρινό πλαίσιο τα χρήματα τα οποία είναι διαθέσιμα για τις μεταφορές θα μπορέσουν να προετοιμάσουν αυτό το πακέτο, την εφαρμογή αυτού του πακέτου επενδύσεων που ανέφερα. Ο Ζωσμπαχ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και καλώς ήρθατε, υποψήφια Επίτροπε. Οι ερωτήσεις μου αφορούν και εμένα τα δικαιώματα των επιβατών και χαιρετίζω τις δηλώσεις και τις απαντήσεις που δώσατε στους προηγούμενους συναδέλφου για την διατροπικότητα και την επιβολή των δικαιωμάτων της ε, προστασίας του σεβασμού των δικαιωμάτων των επιβατών. Πολύ σωστά ξεκινήσατε. Θα ήθελα συγκεκριμένα να ρωτήσω εάν κατά την επεξεργασία των δικαιωμάτων των ε, επιβατών θα θέσετε τον ε, επιβάτη πάντα στο επίκεντρο της προσοχής, γιατί αυτό συνέβαινε πάντα στο παρελθόν. Και επίσης υπάρχει μια σειρά ε, νομοθετημάτων, κυρίως για τις ενέργειες μεταφορές. Συγκεκριμένα η οδηγία 261 Υπάρχουν διαφορές, αποκλίνουσες απόψεις ε, και σε αυτό θα ήθελα να πω ότι λυπούμε που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο δεν έχουν ε, τη δυνατότητα να αναλάβουν ένα κατά κάποιον τρόπο συνταγματικό ε, ρόλο, ένα νομοθετικό ρόλο θα έλεγα. Δεν μπορούσα να ολοκληρώσω το νομοθετικό έργο και έτσι το ζήτημα έμεινε στα χέρια του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για να κρυθεί. Πώς μπορείτε λοιπόν νομίζετε να αντιμετωπίσετε αυτό το αδιέξοδο και να μας βγάλετε από τη το θέμα αυτό του 261 απάντηση. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Συμφωνώ απολύτως ότι αν δεν είναι αρκετά σαφείς οι κανόνες, προφανώς αναγκαστικά ε, παρεμβαίνουν τα δικαστήρια με τις αποφάσεις τους. Οι πρόσφατες δε αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την αποζημίωση στην περίπτωση παραβίασης των κανόνων περί δικαιωμάτων ε, των επιβάτων, αλλά και η απόφαση σχετική με τη δεύτερη χειραποσκευή, όπως ονομάζεται, ε, έχουν μεγάλη σημασία και θα πρέπει να είμαστε πιο σαφείς στην νομοθεσία μας. Εάν προκύπτουν τέτοια ζητήματα δηλαδή θα πρέπει πάντοτε να διευκρινίζονται οι ε, διατάξεις έτσι ώστε και να είναι σεβαστή η νομολογία και οι αποφάσεις του δικαστηρίου αλλά και όπως σωστά αναφέρεται να τεθεί στο επίκεντρο της προσοχής ο επιβάτης. Νομίζω ότι εάν δεν πιέζαμε τόσο για τα δικαιώματα των επιβατών θα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα στις αεροπορικές μεταφορές. Θα είχαμε το overbooking, την ε, κράτηση δηλαδή πλεοναζουσών θέσεων που έχουμε ζήσει όλοι και φτάναμε στο αεροδρόμιο χωρίς να ξέρουμε αν θα μας βάλουμε μέσα στο αεροπλάνο ή όχι ή θα είχαμε άλλου τύπου περιορισμούς που θα δυσκόλευαν πάρα πολύ τη ζωή μας, ιδιαίτερα για όσους ταξιδεύουν με τις οικογένειές τους, με μικρά παιδιά. Αυτό λοιπόν και για να περάσω στο θέμα του Γιβραλτάρ, είναι λυπηρό, λυπηρό το γεγονός ότι χρειάστηκε να παγώσει μεγάλο κομμάτι αυτής της νομοθεσίας και βεβαίω η Επιτροπή έχει υποχρέωση τετερότητα ω προ την ε, κυριαρχία των κρατών μελών. Ε, είμαι διτεθειμένο να συνεργαστώ με εσά και με το Συμβούλιο για να αναζητήσουμε έναν τρόπο να ε, λύσουμε το ζήτημα για να προχωρήσουμε στο νομοθέτημα. Η κυρία Κονσάλης Πένιας, αλλά και πάλι θα, θα παρακαλέσω τον υποψήφιο να τηρεί το χρόνο του. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε η στρατηγική 2020 για την Ευρώπη πρέπει να δημιουργήσει μια περιεκτική και ευφυή και ανταγωνιστική ανάπτυξη. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε όλο και μεγαλύτερη συγκέντρωση αναποτελεσματική των πόρων και επιβολή των συμφερόντων των επενδυτών στο σύνολο της κοινότητας. Και μέσα σε αυτά προκύπτει και όλο μικρότερη υποστήριξη για τις δημόσιες συγκοινωνίες. Αυξάνονται οι αυτοκινητόδομοι, αυξάνονται τα αεροδρόμια τα οποία δεν έχουν κίνηση. Ε, τρένα υψηλής ταχύτητος και δεν είναι όλα αυτά βιώσιμα όπως θα έπρεπε να είναι για την Ευρώπη. Το ερώτημά μου είναι με ποιο τρόπο θα εξασφαλίσετε ότι οι πολιτικές μεταφορών θα χαραχθούν για τους λαούς της Ευρώπης, θα λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες τους και θα λαμβάνουν υπόψη τη σημαντική, σημαντικό ρόλο που έχουν οι μεταφορές για την ευμάρεια και την κοινωνική συμμετοχή και δεν θα ακολουθούν μονάχα τα ιδιωτικά συμφέροντα ορισμένων μεγάλων φορέων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ερώτημά σας. Θέτετε ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό και το οποίο θα έχει μονίμως μεγάλη σημασία στο μέλλον. Αυτό είναι οι δημόσιες μεταφορές. Είναι πολύ σαφές ότι ιδίω τους αστικούς ε, χώρους της πόλης της Ευρώπης δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε με τις τωρινές συνθήκες μεταφορών. Όταν οι επιχειρήσεις μας και οι πολίτες μας χάνουν πάρα πολύ καιρό σε κυκλοφοριακές συμφορήσεις όπου καταστρέφουμε με την ε, ρήπανση της ατμόσφαιρας και την εκπομπή αερίων θερμοκηπίου καταστρέφουμε το περιβάλλον μας και κάνουμε τις πόλεις μας χώρους που δεν είναι ευνοϊκοί για να ζει κανείς. Νομίζω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε προς ε, αηφόρες δημόσιες μεταφορές γιατί αυτή θα είναι μια λύση που θα είναι φιλική προς το περιβάλλον και πιστεύω ότι και οι πολίτες, οι κάτοικοι των πόλεων θα την χαιρετήσουν και με τον τρόπο αυτό θα αντιμετωπιστεί και το θέμα αυτό το οποίο είναι τόσο σημαντικό στην Ευρώπη της απώλειας εκατό του ΑΕΠ μας γιατί τόσες πολλές ώρες κάθε μέρα βρισκόμαστε σε μποτιλιαρίσματα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις ανάγκες των πολιτών, εγώ είμαι έτοιμος να προβούμε σε δημόσιες διαβουλεύσεις με όλους αυτούς οι οποίοι έχουν προτάσεις για να βελτιωθεί η κατάσταση των μεταφορών και ξέρω ότι και με τις πόλεις είμαι έτοιμος να έρθω σε επαφή παρά το γεγονός ότι ξέρω ότι τα κράτη μέλη θα επικαλεστούν την επικουρικότητα και είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε το θέμα της προσβασιμότητας όταν δεν μπορούμε παραδείγματος χάρη να χρησιμοποιήσουμε τους μηχανισμούς αγοράς όπως είναι η επιβολή δημοσίων υποχρέωσεων. Για Ευχαριστώ πολύ. Keith Taylor. Με, με, με τρομάξατε πρόεδρε, νόμιζα ότι δεν ήξερα ποιος είμαι. Κύριε Σεφκοβιτς, με ποια συγκεκριμένα μέτρα θα ενσωματώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το θέμα της δημόσιας υγείας στην πολιτική των μεταφορών, δεδομένου ότι υπάρχουν όλο και περισσότερα επιστημονικά στοιχεία και αποδείξεις ότι προκαλείται καρκίνος, αναπνευστικά νοσήματα, καρδιαγκιακά νοσήματα λόγω των ε, μεταφορών. Και θα ήθελα να συμφωνήσω ότι 26.000 θάνατοι στους δρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαράδεκτα υψηλό νούμερο. Αλλά θα σας καλέσω και εγώ να θυμάστε ότι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε 29.000 νεκρούς το χρόνο από την ατμοσφαιρική ρήπανση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος για την ερώτησή σας νομίζω ότι αποδεικνύεται κατάφορα το πόσο οι μεταφορές είναι αλληλένδετες με τόσους άλλους τομείς πολιτικής και άρα έχουν κρίσιμη σημασία για την ευημερία του Ευρωπαίου πολίτη. Τι μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένα, ρωτάτε, τι μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένα. Νομίζω ότι αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να αναζητήσουμε κάθε δυνατή επιλογή ώστε να μειωθούν ακόμη περισσότερο οι νεκροί από τροχέα στους δρόμους μας. Ήδη, όπως είπα, έχουμε αναλάβει μέτρα. Πρέπει να προχωρήσουμε σε πιο σημαντικά μέτρα, να βελτιώσουμε, να εξεχρονίσουμε τις υποδομές, το φωτισμό των δρόμων, να υποστηρίξουμε τις εξελίξεις αυτές όπου υπάρχει δυνατότητα και με, με ευρωπαϊκά ταμεία. Και πρέπει να δουλέψουμε σε καλύτερους, για καλύτερους στόχους όσον αφορά τους σοφαρούς τραυματισμούς 26.000 νεκροί είναι πολλοί, αλλά και οι 250.000 τραυματίες είναι πολλοί. Ο κύριος Ναι, για την, για την ατμοσφαιρική ρήπανση. Αναφέρθηκα μόλις τώρα στην απάντηση που έδωσα στη συνάδελφό σας η ατμοσφαιρική ρήπανση είναι ένα απαράδεκτο φαινόμενο. Αν δούμε τι συμβαίνει στα αστικά κέντρα και κυρίως τις ώρες της κυκλοφοριακής αιχμής, είναι απαράδεκτη η κατάσταση. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν εδώ. Πώς είπα, πρέπει να φροντίσουμε να σεβαστούμε και τις πολύ λεπτές διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στο αρμοδιότητες τη Επιτροπής των κρατών μελών και των ε, τοπικών ή περιφερειακών αρχών, γιατί θα πρέπει να μπορούν οι, τα αστικά κέντρα να σχεδιάζουν μόνο τους τις μεταφορές όπως τις θέλουν για τον πολίτη του Εγώ είμαι διατεθειμένος να συνεργαστώ και με τις ε, ε, τοπικές περιφερειακές αρχές και με τις κρατικές αρχές, τις εθνικές αρχές για πλατφόρμες δημοσίων μεταφορών, για κινητικότητα καλύτερη, γιατί υπάρχουν πολλές λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πόλεις μας εν γέννη. Ευχαριστώ κυρία Αιούτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητέ κύριε Επίτροπε, ο τομέας των μεταφορών είναι υπεύθυνο του 24% των εκπομπών καυσαερίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι οδικές μεταφορές είναι το 18%. Παρ' όλα αυτά ε, τα οχήματα τα οποία κινούνται με εναλλακτικέ μορφές καυσίμων είναι ελάχιστα. Ε, θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε νέα μέσα όπως ε, οι κινητήρες με πεπιεσμένο αέρα ή οι ε, ηλεκτρικοί κινητήρες. Ή θα συνεχίσουμε να είμαστε όμοιροι των λόμπι των ορυκτών καυσίμων και να απαγορεύουμε σε αυτούς οι οποίοι να προχωρήσουν αυτοί οι οποίοι θέλουν να προωθήσουν νέες καινοτόμες μορφές κίνησης. Θα συνεχίσετε να είσαστε όμοιρος ε, των ε, πολιεθνικών εις βάρος των πολιτών ή θέλετε να κάνετε μία προσπάθεια για να εγκαταλείψουμε τα ορυκτά καύσιμα υπέρ των εναλλακτικών. Μία δεύτερη ερώτηση. Η κυρία Ντελή είχε αναφερθεί στην γραμμή Τωρίνο Λιών και εσείς δεν αναφερθήκατε σε αυτό, την αγνοήσατε. Γνωρίζετε το ότι η γραμμή το Ρήνο ε, είναι μια παραδοσιακή σιδηροδρομική γραμμή και την χάνει Ευρωπαϊκή βοήθεια σαν να ήταν υψηλής ταχύτητας, κάτι το οποίο είναι μια παράνομη χρήση των κοινοτικών πιστώσεων. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, τα εφή e, οχήματα, τα οποία θα κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα. Νομίζω ότι θα πρέπει εδώ ε, να μην μείνουμε σε, στο, ε, σε παραδοσιακού τύπου διλήμματα, εν περιπτώσει, τα οποία είναι αδιέξοδα. Νομίζω ότι ε, δεν υπάρχει, λέγουν ε, κάποιοι οι οποίοι προωθούν τις υποδομές για τα καινοτόμα ε, μέσα, ότι δεν υπάρχει ζήτηση. Πρέπει να προωθήσουμε λοιπόν τα FEE e οχήματα, πρέπει να προωθήσουμε τη χρήση του ηλεκτρισμού για την κίνηση, το υδρογόνο, τις κυψέλες υδρογόνου, πεπιεσμένου αέρα και οι νέες αυτές τεχνολογίες είναι σωστό να προωθηθούν αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τα τέν θα είναι σε θέση να καλυψεί και τις ανάγκες στις καινοτόμες αυτές μορφές κίνησης με εναλλακτικά καύσιμα. Σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι μπορούμε να δούμε περισσότερα ευφυή οχήματα στους δρόμους μας. Ο Γκέορκ Μάιερ. Ως ε, μη εγγεγραμμένος βουλευτής δυστυχώς βρίσκομαι σε μειονεκτική θέση εδώ στο Κοινοβούλιο. Δεν μπορώ να σας υποβάλω ερωτήσεις για επί τρία λεπτά, αλλά μόνο για ένα λεπτό. Αλλά έχω να ρωτήσω το εξή. Ξέρετε ότι η Αυστρία είναι μετά την διεύρυνση προς Ανατολάς το είναι ένα κράτος ε, διέλευσης στις οδικές μεταφορές. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω ε, τι έχετε να προτείνετε για, τις, ε, για τα σχέδια, για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, ειδικά για την Αυστρία και αν, αν υπάρχει δυνατότητα για πραγματική χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα Ευρωπαϊκά κόνδυλα. Και μια πρόκειται για κράτος ε, διαμετακόμισης, ε, διέλευσης. Δεν θέλω να ρωτήσω αν σκοπεύετε να κάνετε κάτι για τα πολύ παλιά φορτηγά ε, που κυκλοφορούν στους δρόμους της Ευρώπης, τα οποία αποτελούν κίνδυνο για τους πάντες. Τι θα κάνετε γι' αυτό λοιπόν. If I may ask you, Εάν ε, μου επιτρέπετε η ερώτησή σας αφορά συγκεκριμένα την σύραγγα στην Αυστρία ή, ή Όχι, έχουμε δύο. Το COARM και το Σαν Μαρίν. Οι δύο αυτές σύραγγες με ενδιαφέρουν. Ναι, ευχαριστώ. Νομίζω ότι αυτό πάλι σχετίζεται με, την με τις προηγούμενες ερωτήσεις και το θέμα των ε, σειραγγών στους δρόμους. Ξέρετε ότι είναι πολύ δύσκολη και περίπλοκη συζήτηση για τα TNT, για τα, για τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα δηλαδή Μεταφορών. Επίσης γνωρίζετε ότι όλοι μας, Συμβούλιο, Κοινοβούλιο και Επιτροπή, συμφωνήσαμε ότι εφόσον θέλουμε αυτή η θετική μετακύληση να πραγματοποιηθεί με πραγματική αλλαγή στις υποδομές στην Ευρώπη θα πρέπει να εστιάσουμε τα μέσα, τα κονδύλια που έχουμε στη θέσή μας σε πραγματικά έργα που θα οδηγήσουν σε ουσιαστικές βελτιώσεις στις υποδομές. Εξού και η επιλογή να ακολουθούν συμφωνημένα ε, έργα, μεθοδολογία, με διεξοδική συζήτηση που θα ε, ενέκρινε πρώτα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι για μένα κάθε ένα από αυτά τα έργα είναι ισοδύναμο με νομοθεσία ευρωπαϊκή, γιατί το έχετε εγκρίνει εσείς. Πλέον έχει μείνει μόνο η εκτέλεση των έργων που έχετε ε, ψηφίσει και εγκρίνει. Έτσι θα χειριστώ οδήποτε από αυτά τα έργα των διευρωπαϊκών δικτύων. Τώρα για να περάσω στο θέμα των ε, φορτηγών. Νομίζω ότι θα χρειαστώ περισσότερο από τα δευτερόλεπτα που μου λείπουν για τα πολύ μεγάλα φορτηγά, αλλά μια και ο πρόεδρος είναι τόσο ευστηρός με τον χρόνο, θα πρέπει να περιμένω την επόμενη ερώτηση. Ευχαριστώ κυρία Κριστίν Ρεβόντα Λόν Μπονφουά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε το σιδηρομικό πακέτο να, να συζητηθεί στο σύνολό του. Αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχει κίνδυνος ε, να μην καταλήξουμε κάπου. Θα εγκαταλείψετε σε αυτή την περίπτωση τις προσπάθειες για την τεχνική συμφωνία. Για τη συμφωνία στα τεχνικά θέματα πάνω στα οποία έχει γίνει πολλή δουλειά και έχουν βρεθεί και κοινή Τώρα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ε, Σιδηροδρόμων, η οποία μειώθηκε ο προϋπολογισμός, οποίας μειώθηκε ο προϋπολογισμός κατά 5%. Αυτό πώς επηρεάζει το τεχνικό κομμάτι, πώς προβλέπετε εσείς να λειτουργήσει η υπηρεσία αυτή με περισσότερες αρμοδιότητες και μικρότερο προϋπολογισμό. Σας ευχαριστώ κυρία σχετικά με τις εξωτερικές υπηρεσίες πράγματι μου ξανάρχονται αυτά από το παρελθόν. Ήμουν υπεύθυνο για τις ε, διαπραγματεύσεις των νέων αυτών ρυθμίσεων ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις εξωτερικές υπηρεσίες. Πάντως είναι σαφές ότι η υπηρεσία συνδρομική η ευρωπαϊκή είναι στην φάση οικοδόμησης, δημιουργίας και ολοκλήρωσης και είναι μια υπηρεσία για το μέλλον. Εγώ θα ανέμενα, αν θυμάμαι καλά, 43 επιπλέον θέσεις προσωπικού να δοθούν στην υπηρεσία αυτή, ε, που σε κάποια φάση θα αυξήσουν το προσωπικό τους γύρω στα 200 άτομα. Είναι σημαντική αύξηση αυτή. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό σε ένα ευρύτερο κλίμα μειώσεων 5% ε, στο σύνολο των εξωτερικών θεσμικών οργάνων και υπηρεσιών. μπορούμε να το πετύχουμε μέσω της χρηματοδότησης ε, των νέων εμπειρογνωμόνων που οργάζονται για την συγκεκριμένη υπηρεσία μέσω των ανταποδοτικών τελών. Ξέρετε ότι θα χρεώνουν για τις αδειοδοτικές τους ε, δραστηριότητες. Η υπηρεσία αυτή ε, είναι κάτι το οποίο αναμένεται ιδιαίτερος από την βιομηχανία της ηροδρομική θέλουν να, να απαλλαγούν από τις 26.000 εθνικούς κανόνες που εφαρμόζονται σήμερα και να μειώσουν και τον χρόνο αδειοδότησης νέων, νέου υλικού σιδηροδρομικού, τροχαίου υλικού και πρέπει να περνάει από εθνικές υπηρεσίες πολλαπλές ενώ τώρα τα πράγματα θα πηγαίνουν πολύ πιο γρήγορα και η τεκμηρίωση θα είναι ταυτόσιμη σε όλα τα κράτη-μέλη. Λοιπόν, τα χρήματα που θα δαπανίσουν οι υπηρεσίες αυτές θα είναι χρήματα τα οποία θα δαπανηθούν σωστά και έτσι θα καλύψουμε την αύξηση του προσωπικού. Και τώρα περνάμε στις ερωτήσεις από την Επιτροπή Ήτρε και καλωσορίζω τον πρόεδρό της, κύριο Μπούζεκ. Η κυρία Νίμπλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Κύριε υποψήφι, επίτροπε, από τις μεταφορές πάμε στο διάστημα και έχω ερώτηση για το Γαλιλαίος. Είναι ένα από τα ε, μεγαλειώδη εγχειρήματα της Ευρώπης που έχει υποστηριχθεί ανέκαθεν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και θέλω να σας ρωτήσω, εφόσον επιβεβαιωθείτε ε, στον τουρισμό αυτόν, θα συνεχίσετε με, την ίδια, ε, με τον ίδιο ενθουσιασμό στο έργο αυτό του Γαλιλαίου όπως και προκατοχό σας και επίσης για την ανάπτυξη του Γαλιλαίου έχετε πει ε, από την αρχή ότι σας ενδιαφέρει το θέμα των δορυφόρων, αλλά είχαμε προβλήματα στην εκτόξευση των δύο τελευταίων δορυφόρων. Θα γίνει λοιπόν κάτι. Επίσης για το θέμα των ε, διπλωμάτων ευρεσιτεχνία και τη του τοκτησία στο Γαλλέο, γιατί ασφαλώ θα χρειάζεται κάποιο είδου αδειοδότηση για την πρόσβαση στα δεδομένα. Επίση, ε, η χρήση τόσο εμπορική όσο και από κρατικέ δημόσιε υπηρεσίε για το Γαριλαίο. Θα με ενδιαφέρει να μου πείτε τι σκοπεύετε να κάνετε γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Νιμπλερ. Για την πρώτη σας ερώτηση, απερίφραστα ναι διότι έχουμε εργαστεί για τόσα χρόνια με το ε, εγχείρημα αυτό του Γαλιλαίου. Ο προκάτοχος μου κ. Σταλιάν ήταν αυτός ο οποίος τακτοποίησε τα του Γαλιλαίου. Έχουμε μια καλή ομάδα που δουλεύει για το έργο αυτό. Έχουμε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για το τι θέλουμε να κάνουμε. Και αυτή τη στιγμή νομίζω, γιατί σήμερα έγινε ακόμη μια ε, έρευνα ε, μια συνάντηση στην ε, Μόσχα, μια συζήτηση στη Μόσχα που ήθελε να διερευνήσει ακριβώς ποια ήταν τα προβλήματα, γιατί, γιατί εμφανίστηκε αυτό το injection anomaly, αυτό το πρόβλημα έγχυσης και πώς μπορούμε να σώσουμε τους δορυφόρους, γιατί αν δεν μπορέσουμε να τους αξιοποιήσουμε, καλό θα είναι τουλάχιστον να μην τους χάσουμε τελείως, ακόμα και βρεθούν σε διαφορετική τροχιά, θα πρέπει να μπορούμε να αξιοποιήσουμε την παρουσία τους στο διάστημα, αλλά πάλι εδώ θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε ουσιαστικά αποτελέσματα από την έρευνα αυτή, από την Επιτροπή Έρευνας. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε εάν μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα του, της θέσης σε τροχιά, αν μπορεί να αντιμετωπιστεί δηλαδή το ε, ολίσθημα αυτό ε, ή, εν πάση περιπτώσει, για να είμαι και πιο σαφής, εγώ θα ήθελα να διαρευνηθούν διεξοδικά όλα τα τεχνικά προβλήματα που ενδεχομένω εμφανίζονται για να είμαστε σίγουροι ότι αναπτύσσεται σωστά το έργο. Ε, στη συνέχεια θα πρέπει να έχουμε την, το REN5 με τον τέταρτο δορυφόρο και άρα θα μπορεί το έργο Γαλιλαίος να αναπτύχθει σε, σε αυτό το στερέωμα που ονομάζεται Daily Service. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Σεύκοβιτς, σας χαιρετίζω και σας καλωσορίζω για την παρουσία σας. Καταρχήν, είχα την ευκαιρία να δω το έργο σας στην τωρινή θητεία της Κομισιόν Δείξατε ενεργητικότητα και μεγάλη αποτελεσματικότητα. Σας εύχομαι να συνεχίσετε και στην επόμενη Επιτροπή. Είδα να έχετε ένα σαφές όραμα σε σχέση με την ανάπτυξη των θεμάτων στο χαρτοφυλακείό σας που είναι εκτενές και πολύπλοκο, έχει πολλές δυνατότητες. Θα ήθελα όμως να σας θέσω ένα ερώτημα πιο συγκεκριμένο. Ποια είναι η άποψή σας για την διαστημική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ποιες είναι οι κέρδιες πρωτοβουλίες που έχετε σαν στόχο να ξεκινήσετε έχετε την πρόθεση να παρουσιάσετε μια πολιτική για εκτοξευτές ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ανεξάρτητη πρόσβαση στο διάστημα λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό μπορεί να είναι από τα κυριότερα προβλήματα που θα συζητηθούν το Δεκέμβριο στη συνάντηση Ευρωπαϊκής Ένωσης Πολιτειών. Ποια άλλα μέτρα επίσης θα λάβετε στον τομέα της εξερεύνησης του διαστήματος που είναι ένας από τους κύριους στόχους της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Διαστήματος. Σας ευχαριστώ πολύ <clears throat> για τα θερμά σας λόγια, αλλά νομίζω ότι η ενεργητικότητα και η αποτελεσματικότητα είναι κέρια στοιχεία για την διαστημική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τα θέματα μεταφορών ισχύει αυτό, αλλά ισχύει και για τη διαστημική μας πολιτική. Έχουμε μπροστά μας, τα έλεγα, τα πιο κέρια πέντε χρόνια για την ευρωπαϊκή διαστημική πολιτική πιο σημαντικά από ό,τι ποτέ. Θέλουμε ο Γαλιλαίος να φτάσει στην πλήρη ανάπτυξή του. Δηλαδή σχεδόν 30 δορυφόρους, εξαρτάται πόσοι από αυτούς θα είναι σε τροχιά και ποιοι, πόσοι θα είναι σαν δορυφόροι ε, ενδεχόμενης αντικατάστασης. Επίσης θέλουμε να πράξουμε το ίδιο και με το πρόγραμμα Κοπέρνικος, όπου θέλουμε να αναπτύξουμε 12 δορυφόρους παρακολούθησης της γης, γιατί ο Γαλιλαίος είναι περισσότερο για το σύστημα ε, εντοπισμού και επίσης και για την ε, διατήρηση της ακρίβειας των ατομικών ρολογιών, ώστε παραγωγικά να γίνεται σαφής η χρονική στιγμή των ε, συναλλαγών που γίνονται σε χρηματοπιστωτικά ανταλλακτήρια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν η Ευρώπη να εξασφαλίσει την ε, ανεξαρτησία της και όχι να βγει από το παιχνίδι μόνο και μόνο επειδή δεν έχουμε την αυτόνομη πολιτική διαστήματός μας. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τους εκτοξευτές υπάρχουν ε, αναλύσεις που έχουν γίνει και προπαρασκευαστική εργασία για το πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε την Αριάν 5 ή την Αριάν 6 και έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν θα έχουμε μονάχα ένα μεγάλο εκτοξευτή όπως είναι η Αριάν 5 και ένα μικρό εκτοξευτή όπως είναι το Ρέγκαν, αλλά και κάποιον ενδιάμεσο για τις ε, ε, εκτοξεύσεις που γίνονται από ξένους πυράβλους αυτή τη στιγμή. Λουτουλόφσκι. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η υποψηφία επίτροπε. Θα μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα για να σας ρωτήσω για την πολιτική του διαστήματος που αφορά τις αρμοδιότητες της Επιτροπής ΣΥΤΡΕ. θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο το σύστημα δορυφορικής πλοήγησης ε, που θα αναπτυχθεί με το έργο Γαλιλαίος. Πιστεύετε ότι μπορούν να υπάρχουν συνεργατικές σχέσεις και να αναλάβει με τον τρόπο αυτόν η νέα υπηρεσία ε, νέα καθήκοντα όπως με το Κοπέρνικος αλλά και με αντίστοιχα άλλα ε, έργα τα οποία από μόνα τους θα μπορούσαν να φανούν είτε πολύ δαπανηρά είτε και περιτά. Ευχαριστώ πολύ και χαίρομαι που μπορώ να σας απαντήσω στην ε, μητρική μου γλώσσα τώρα γιατί ξέρω ότι θα με καταλάβετε αν μιλάω σλοβακικά. Για το μέλλον λοιπόν και την ε, υπηρεσία αυτή της πράγας. Μπορεί να πει κανείς ότι έχουμε εδώ αναπτύξει προτεραιότητες για το μέλλον με την ε, υπηρεσία αυτή και το γεγονός ότι ξεκινάει αυτή η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα να ε, αξιοποιηθεί και εμπορικά ο Γαλιλαίος. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν το ε, ε, έργο αυτό για τον Ευρωπαίο πολίτη αλλά και για την επιχείρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει ευρύτατα καθήκοντα να επιτελέσει. Εδώ μιλήσαμε για το Κοπέρνικο νωρίτερα. Πάνω από 100 αεροδρόμια της Ευρώπης αξιοποιούν το σύστημα αυτό διότι είναι πολύ πιο φθηνή η τεχνολογία αυτή και πολύ πιο σύγχρονη. Επίσης είμαι πεπισμένος ότι η χρήση και αξιολόγηση, αξιοποίηση στοιχείων που μπορούμε να αντλήσουμε από το σύστημα Κοπέρνικος θα πρέπει να ε, γίνει κατά τρόπον ώστε οι πληροφορίε να αξιοποιούνται στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Με την προετοιμασία που έκανα για τη σημερινή ακρόαση, διαπιστώνω ότι τα δεδομένα του Κοπέρνικου σημαίνουν πάρα πολύ ουσιαστική δουλειά ε, στην, για να είμαι ακριβής σημαίνουν νούμερα της τάξης του 1 στην ε, του 1 με 15 μηδενικά, γιατί δεν μπορώ να σας διαβάσω το νούμερο, ε, και άρα τα δεδομένα αυτά σημαίνουν τεράστιες δυνατότητες και για την Επιτροπή, πληροφορίες που μπορούν να αξιοποιηθούν, πληροφορίες μπορεί να χρησιμοποιήσει η Frontex ή κάποιες άλλες υπηρεσίες όπως η περιβαλλοντική, η υπηρεσία, η υπηρεσία για την ασφάλεια στις τεράστιες μεταφορές. Δηλαδή έχει τεράστιο δυναμικό για εφαρμογές. Ευχαριστώ ο κύριος Κρικέ, ο οποίος κάθεται και πίσω σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Υποψήφιοι Επίτροπε, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση για το διάστημα, μια και είναι η σειρά του, αλλά και ως Αντιπρόεδρος Επιτροπής των Μεταφορών για τις μεταφορές. Για το διάστημα Υπάρχει μια πρόταση για υποστήριξη βιομηχανική των χερσαίων εφαρμογών του Γαλιλαίου. Αυτό έχει γίνει με την προηγούμενη Επιτροπή. Αυτό υπάρχει σε επίπεδο, σε στάδιο προετοιμασίας και αφορά ύψους αρκετών δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση και δεύτερον σκοπεύετε να υποστηρίξετε περισσότερο τις δυνατότητες εκτόξευσης και κυρίως βαρέως βε, βαρέως ε, επίπεδου. Και επίσης θα ήθελα να ρωτήσω ε, για τις οδικές μεταφορές και για τις μεταφορές γενικότερα και τους ε, αποσπασμένους εργαζομένους που να λάβετε κάποια μέτρα. Για τις οδικές μεταφορές έχετε κάτι επιπλέον να μας πείτε για την ασφάλεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ρικέ. Κύριε Αντιπρόεδρε. Θα πρέπει να βελτιώσουμε την αποδοχή από τον επιχειρηματικό κόσμο του Γαλιλαίου στο βαθμό που μπορούμε και όπου μπορούμε πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει ώστε να υπάρξουν νέες αποδέκτες για το σύστημα και να είναι ε, συμβατά τα συστήματα όπως το οίκο παραδείγματι με το Γαλιλαίο. Σε όλος ο εξοπλισμός ο οποίος σχετίζεται με την έρευνα και διάσωση στις διάφορες, τις διάφορες περιοχές κρίσης, όπου έχουμε σαφέστατες ρυθμιστικές εξουσίες, μπορούμε να επιβάλλουμε, να είναι συμβατός ο εξοπλισμός με το Γαλιλαίο. Επίσης πιστεύω ότι πρέπει να εργαστούμε στενά σε συνεργασία και με τον κλάδο και με τις υπηρεσίες ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι όταν ε, αρχίσει να εκπέμπει σήμα ο Γαλιλαίος θα έχει ε, μαζική αποδοχή και θα φέρει τους καρπούς του απευθείας στον, ε, στην οικονομία της Ευρώπης, επιχειρήσεις της Ευρώπης, γιατί θα είναι πολύ πιο ακριβής ο Γαλιλαίος θα έχει δίνει δηλαδή πολύ πιο ακριβή στοιχεία αναγνωρίσιμα από ό,τι γνωρίσουμε τώρα από το σύστημα GPS και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε οτιδήποτε περνάει από το χέρι μας. Ε, λαμβάνονται όμως και όλα τα μέτρα, αναλαμβάνονται όμως και όλα τα μέτρα για την ορθή εφαρμογή του Γαλλιού. Για τους εκτοξευτές ε, είναι μεγάλου βεληνικού έργου, έργο, αλλά βεβαίως ε, τάσσομαι υπέρ ιασδήποτε επιλογής που θα μας εξασφάλιζε αυτονομία στο διάστημα. Ευχαριστώ, επόμενος μιλητής. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να δώσω τη δυνατότητα στον κύριο υποψήφιο επίτροπο να μιλήσει σλοβάκικα και γι' αυτό θα θέσω ένα ερώτημα στα τσεχικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα να αναφερθεί ο κύριος Επίτροπος για τα θέματα θαλασσίων μεταφορών και εσωτερικών υδατίνων δρόμων ε, που χρησιμοποιούνται μόνο σε περιορισμένο επίπεδο 15% σε ορισμένε περιπτώσει. Τι θα κάνετε λοιπόν για άλλους ποταμούς, τι θέλετε να κάνετε. Στην Λευκορωσία θέλουν να συνθέσουν τον δυτικό Δβίνα στον Δνήπερο, κάτι το οποίο θα επιταχύνει τις ε, διελεύσεις κατά τέσσερις φορές από τη Μεσόγειο στην Βαλτική θάλασσα. Θα ήθελα να ξέρω αν θέλετε να υποστηρίξετε το φιλόδοξο σχέδιο του πρόεδρου μας, του Μίλο Ζέμαν, σύνδεσης μεταξύ ε, Δούναβη και Όντερ και Έλβα. Με τη σύνδεση λοιπόν αυτή θα, έχουμε, θα υπάρχει σύνδεση τριών ευρωπαϊκών ε, θαλασσών, αλλά με τον τρόπο αυτό θα παραβιαστεί και η γερμανική νομοθεσία γιατί το Βραδεμβούργο και η Σαξονία έχουν ήδη βγάλει ένα κοινοβουλευτικό ψήφισμα για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ, λέει ο κύριο ε, Σεύκοβιτς. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να μιλήσω την μητρική μου γλώσσα και να σας ευχαριστήσω για το ερώτημά σας που δείχνει και πάλι τη σημασία του να χρησιμοποιήσουμε το δυναμικό το οποίο υπάρχει στις εσωτερικές πλωτές μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αυτή τη στιγμή δεν έχει χρησιμοποιηθεί πλήρως. Οι δυνατότητες λοιπόν οι οποίες υπάρχουν σε αυτό το τομέα είναι φυσικά περιορισμένες λόγω του προϋπολογισμού μας αλλά χαίρομαι και για την υποστήριξη που έχω λάβει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μας έδωσε το ίδιο επίπεδο πόρων όπως και στην προηγούμενη θητεία, στην προηγούμενη δημοσιονομική περίοδο μάλλον, και με τον τρόπο αυτό μπορούμε να υποστηρίξουμε σχέδια για εσωτερικές διαδρομές στον Δούναβη, μπορεί να ανανεωθεί ο στόλος των ποταμοπλοίων, γιατί υπάρχουν πολλά από αυτά τα οποία είναι πεπαλαιωμένα. <clears throat> μπορούμε επίσης να βελτιώσουμε τις λιμανικές υποδομές και των, ε, τις υποδομές των καναλιών στις παραδυνάβιες περιοχές. Μας ενδιαφέρει όμως να προχωρήσουμε και σε καλύτερη κατάρτιση του, των εργαζομένων στις εσωτερικές υδάτινες διαδρομές. Πολλές φορές και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο σε αυτό το τομέα. Για τα σχέδια που ανέφερε ο κύριος βουλευτής, το ερώτημα είναι πώς θα μπορούσε να εξασφαλιστεί ότι είναι συμβατά με τα τέντη και με τις χρηματοδοτικές δυνατότητες που έχουμε στον τομέα αυτό. Ο κύριος Κόμπορν, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε υποψήφια επίτροπε, θα συμφωνούσατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίω στον τομέα μεταφορών, δεν θα πρέπει να κατασπαταλά τα χρήματα των φορολογουμένων σε προγράμματα υψηλού κύρους που δεν ευνοούν και δεν ωφελούν κανένα από τους ε, φορολογούμενους. και το τελευταίο τέτοιο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην Νότια Ευρώπη. Συμφωνείτε ότι αυτά τα σχέδια μεταφορών είναι και αυτά ένα είδος φαντασιώσεως να, που έχει σαν στόχο να μιμηθούμε τους Αμερικανούς. Το πρόγραμμα Γαλιλαίος και Κοπάνικος δεν έχει καμία σχέση με τις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών και των Βρετανών υπηκόων. Το να μπορεί κανείς να εξασφαλίζει ότι μπορεί να φορολογεί όλα τα αυτοκίνητα των Ευρωπαίων όταν κινούνται στην Ευρώπη. Αυτός είναι ο στόχος, ενώ υπάρχει μια λιτότητα που καλύπτει όλους. Θα χρησιμοποιήσετε τη θέση σας να σταματήσετε αυτό το παράλογο, το μεγαλόσχημο σχέδιο το οποίο είναι σε βάρος των φορολογουμένων. Σίγουρα η ιδιωτική αγορά είναι σε πιο καλή θέση για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της διαστημικής βιομηχανίας από ό,τι κράτη ή η νομενκλατούρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως υποψήφιος επίτροπος θα πρέπει να σας ευχαριστήσω και για αυτό το ερώτημα. Κατανοώ βέβαια ότι εδώ φαίνουμε απόψεις που θα έπρεπε να περιληφθούν στη συζήτηση. Πιστεύω όμως και από την προηγούμενη δήλωσή μου θα έχετε κατανοήσει ότι δεν συμμερίζομαι με, με τις απόψεις που έχετε εκφράσει για την ευρωπαϊκή πολιτική διαστήματος και φυσικά δεν συμφωνώ και με την περιγραφή που έχετε δώσει για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα ευρωπαϊκά κονδύλια στον τομέα αυτό. Γιατί είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι η Ευρώπη χρειάζεται ένα διαστημικό πρόγραμμα. Χρειαζόμαστε την ανεξαρτησία μας στον τομέα αυτό και την αυτονομία μας σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στο διάστημα και δεν είναι μονάχα θέμα κύρους, μονάχα και ακτινοβολίας. Δεν είναι θέμα κύρους, δεν είναι θέμα ακτινοβολίας. Το χρειαζόμαστε για την τεχνολογία μας ε, εχμής, για τα ευφύ συστήματα μεταφορών, για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα συμφόρησης της πόλης μας. Τα χρειαζόμαστε και για τον τραπεζικό μας τομέα ακόμα. Αν ρωτήσετε τους συναδέλφους σας στο City του Λονδίνου, θα σας πούν πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει η σφραγίδα των ατομικών ορολογίων για όλες τις συναλλαγές που γίνονται στο City του Λονδίνου. Δεν θα πρέπει εδώ να εξαρτιόμαστε μονάχα σε ένα σύστημα όσο καλό και να είναι. Εμείς συνεργαζόμαστε φυσικά με το GPS, αλλά πιστεύω ότι η Ευρώπη είναι αρκετά όρημη, αρκετά ανεπτυγμένη για να έχει τα δικά της συστήματα τα οποία από ό,τι γνωρίζω υποστηρίζονται και από τους Αμερικανούς εταίρους μας. Ευχαριστώ. Jetzt hat das Wort έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ. Όχι, ε, θέλω να επισημάνω ότι πάλι εδώ έχουμε τις ερωτήσεις Επιτροπή Σίτρε και θέλω να ευχαριστώ τον Πρόεδρο και δίνω το λόγο στην ε, κυρία Σμιτ. Ευχαριστώ πολύ ένα ενιαίο οικονομικό και νοσηματικό χώρο απαιτεί και ενιαίο χώρο των μεταφορών. Ωστόσο, στην χρονική στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν 23 διαφορετικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με το, η συζήτηση για την επιβολή διοδίων στου γερμανικού δρόμου ανοίγει ένα μεγάλο κεφάλαιο. Θα Εάν λοιπόν ελοποιηθούν τα σχέδια της Γερμανίας, λαϊκιστές και σε άλλες χώρες της Ευρώπης θα, χρειαστεί, θα θελήσουν να εφαρμόσουν αντίστοιχα συστήματα, πράγμα το οποίο οδηγεί σε δυσφορία, σε αισθήματα ε, δυσάρεστα και βέβαια οδηγεί και στον κατακαιρματισμό των μεταφορών και στον παραλογισμό τελικά. Εδώ δεν μπορούμε να έχουμε δηλαδή ένα ενιαίο χώρο των μεταφορών. Δεν είναι δυνατόν τα εθνικά κράτη να κάνουν διακρίσεις ε, και αυτό να γίνεται ανεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ρωτώ λοιπόν πώς στάσεστε σε περίπτωση επιβολής ενός ε, συστήματος επιβολής διοδίων κατά τρόπο ε, που επιβάλλει διακρίσεις. Σκοπεύετε να αναλάβετε δράση σε μελλοντική συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών της Γερμανίας. Ο πρόεδρος, νομίζω ότι πάλι και εσεί θα πρέπει να δώσετε μόνο σα την απάντηση για να αφήσετε χρόνο στον ερωτόμενο. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω ότι στην Ευρώπη έχουμε και κάποια προβλήματα. Έχουμε... Είμαστε καλοί στη δημιουργία υποδομών, αλλά δεν είμαστε πολύ καλοί στην συντήρησή τους επενδύουμε πάρα πολλά χρήματα για δημιουργία υποδομών αλλά δεν έχουμε την δυνατότητα προσέλκυσης ε, επενδύσεων για τη συντήρηση των υποδομών αυτών. Ε, γι' αυτό ακριβώς ε, ε, το τι θα γίνει με τα εξωτερικά κόστη και πόσο μπορεί να καλυφθούν αυτό είναι κάτι το οποίο δείχνει ότι θα πρέπει να είμαστε ικανοί να βρούμε πηγές χρηματοδότησης οι οποίες ε, να καλύπτονται και φυσικά από τους χρήστες των υποδομών σε σχέση με την ποσότητα βέβαια ε, και το ποσοστό χρήσης τους. Όταν διασχίζει κανείς την Ευρώπη με αυτοκίνητο και πληρώνει διόδια και στο τέλος βλέπει κανείς ότι δεν μπορεί να διακρίνει πολύ εύκολα προς τα έξω γιατί το παμπρίζ του έχει καλυφθεί από όλες τις βινιέτες που πληρώνει ε, υποχρεωτικά στις χώρες τις οποίες διασχίζει. Λοιπόν, το σύστημα θα πρέπει να γίνει πιο δίκαιο, ιδιαίτερα σε σχέση με τον χρόνο χρήσης των υποδομών. Υπάρχει δυνατότητα η τεχνολογική και φυσικά η αρχή της έλλειψης διακρίσεων ε, είναι στη συνθήκη, είναι μια αρχή την οποία σέβομαι και θα σέβομαι. Λιμπεράτσκι έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η πρώτη μου ερώτηση είναι η εξής. Έχουμε ένα νέο μέσο, τον μηχανισμό για τη διασύνδεση στην Ευρώπη, που θα μας επιτρέψει να επενδύσουμε και στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την ισορροπία ανάμεσα στους σιδηροδρόμους και στις οδικές μεταφορές. Στη χώρα μου επιμένουμε κυρίως στις δεύτερες. Ε, θα πρέπει να μιλήσουμε για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και των δύο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε επίσης και τα προγραμματικά ομόλογα, τα project bonds, για να χρηματοδοτήσουμε επίσης και τους μηχανισμούς διασύνδεσης στην Ευρώπη. Ε, μία άλλη ερώτηση. Θα πρέπει να υπάρξει ένας επίτροπος ο οποίος στην ουσία να καταστεί αυτό που θα ονόμαζα ένας υπουργός μεταφορών, όχι μόνο κάποιος που θα σχεδιάζει. Έχουμε τα προβλήματα με το ρωσικό εμπάργκο, αυτό δεν θίγει μόνο ε, τους παραγωγούς οποροκυπευτικών και γαλακτοκομικών αλλά και τους μεταφορείς οι οποίοι μετέφεραν ακριβώς αυτά τα προϊόντα. Ε, θα ασχοληθείτε με το θέμα αυτό. Όταν αναφερθείτε στα, στα θέματα των σχέσεων με την Ρωσία θα παίξετε τον ρόλο του Υπουργού Μεταφορών Είδαμε επίσης το τι κάνει η Γαλλία σε σχέση με το χρόνο ανάπαυσης ε, των οδηγών φορτηγών. Ε, νομίζω ότι είναι κάποιες ιδέες οι οποίες ε, θα άρεσαν και σε μένα και σε εσάς. Κοιτάξτε, λέει ο κ. Σεύκοβιτς, για την διασφάλιση της σωστής ισορροπίας ανάμεσα στα διάφορα TNT. Νομίζω ότι έχουμε συμφωνήσει και στο Κοινοβούλιο για το ποια θα είναι η μεθοδολογία την οποία θα ακολουθήσουμε και τι κατανομή θα υπάρξει στον τομέα της χρηματοδότησης. Ένα ποσοστό δηλαδή της κάλυψης ε, της χρηματοδότησης ε, του Connecting Europe θα αφορά τις περιοχές οι οποίες υπάρχουν προβλήματα για το πέρασμα από τη μια χώρα στην άλλη και γενικά θα ασχοληθεί με τις αιστείες των προβλημάτων των ευρωπαϊκών μεταφορών. Ε, στην περίπτωση τώρα των προγραμματικών ομολόγων, νομίζω ότι σαν μέλος της Επιτροπής Μπαρόζο 2, εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε ένα καλύτερο τρόπο χρήσης τους και να προσπαθήσουμε να βρούμε και άλλους καινοτόμου τρόπους προσέλκυσης των ιδιωτικών επενδύσεων στις ε, υποδομές και στην ανάπτυξη των υποδομών. Σε σχέση με το ρωσικό εμπάργο είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί στα πλαίσια του νέου συνόλου των επιτρόπων και θα προσπαθήσω να εκφραστώ πάνω σε αυτό και στις επαφές που θα έχουμε με τους Ρώσους εταίρους. Πεις επόμενος. Äh, Az a 9 eh, TNT Ένα από εννέα, ένας από τους νέους, από τους εννέα διαδρόμους των TNT είναι αυτός που συνδέει το Ρήνο με τον Δούναβη και θα είναι μια από τις σημαντικότερες συνδέσεις ανατολικά από τα ανατολικά προς τα δυτικά στην κεντρική Ευρώπη, από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι τον ε, Ρήνο. Αυτό είναι τμήμα μια στρατηγική για το Δούναβι τη Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει σαν στόχο να προωθήσει την κινητικότητα και διατροπικότητα στου εσωτερικού υδάτινου δρόμου. Αλλά η ευρωπαϊκή διάτινη δρόμη δεν είναι μονάχα σημαντική για τα κράτη-μέλη, αλλά και για τα συνδυόμενα με την Ευρωπαϊκή Ένωση κράτη όπως είναι η Σερβία, η Βοσνία Ζεγοβίνα, η Μολδαβία, η Ουκρανία. Με ποιο τρόπο έχετε την πρόθεση να εξασφαλίσετε υποψήφια επίτροπε ότι αυτές οι μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες θα έχουν και αυτές την χρηματοδοτική ικανότητα να εφαρμόσουν σχέδια τα οποία είναι κέρια και αυτά για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών υδάτινων δρόμων. Σας ευχαριστώ πολύ για το ερώτημά σας. Έχετε μεγάλο δίκιο ότι ο διάδρομος Ρήνου Δούναβη θα είναι πολύ σημαντικός. Σας ευχαριστώ επίσης και για το ενδιαφέρον σας σε σχέση με χώρες όπως η Σερβία, η Μολδαβία, η Βοσνία Ζεγοβίνη. Πρέπει να πω <clears throat> ότι ενθαρρύνθηκα πάρα πολύ όταν είδα ότι οι χώρες αυτές ενδιαφέρονται και έχουν ενθουσιασμό για τη στρατηγική του δύναμη. Ήταν μία από τις πρώτες μακροστρατηγικές που αναπτύχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την περιοχή του Δούναβη και νομίζω ότι τα, η ελκυστικότητα αυτής της στρατηγικής είναι ότι χάρη στην συνολική αντιμετώπιση που είχε η Κομισιόν που καλύπτει κράτη-μέλη και γειτονικά κράτη μπορούμε να επιτύχουμε πολύ καλύτερη συνέργεια μεταξύ των διαφορετικών εργαλείων χρηματοδότησης και των ταμείων για να έχουμε σχέδια τα οποία είναι πιο ολοκληρωμένα με καλύτερη σύνδεση και μπορούν να φέρουν μεγαλύτερη προσθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή είναι μια προσέγγιση λοιπόν που εγώ θα ήθελα να την υποστηρίξω ιδιαίτερα και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι πάρα πολύ σαφές ότι η πρώτη μας προτεραιότητα και η κύρια εστίασή μας είναι να επιτύχουμε πρόοδο στα θέματα αυτά και εν καιρό να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε την ανάπτυξη ενός διευρωπαϊκού δικτύου για υδάτινους δρόμους. Ξέρουμε όμως ότι αυτοί οι δρόμοι δεν σταματάνε στα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τη συνέχιση τους και σε γειτονικέ χώρες. Αυτό θα είναι και ευνοϊκό για τους Ευρωπαίους πολίτες και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις γιατί έτσι μπορούν να μεταλαμπαδεύσουν τη γνώση, την εμπειρία, το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας με τους γείτονές μας. Είναι καλό για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις. Η Βίκη Μέιερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω τρεις συγκεκριμένες νομίζω ερωτήσεις. Πρώτον, ε, για το φιάσκο του, προηγούμενου μήνα. Εγώ δεν είμαι στην Επιτροπή Θα ήθελα να μάθω όμως ε, ποιες θα είναι οι συνέπειες από την αποτυχία ε, της, της θέσης τροχιά των δύο ε, δορυφόρων και τι θα κοστίσει στους φορολογούμενους. Δεύτερον, με ποιο τρόπο θα μειώσετε την γραφειοκρατία στον τομέα των μεταφορών. Και τρίτον, κύριε υποψήφιε επίτροπε, τι θα κάνετε με τις κίτρινες κάρτες των κοινοβουλίων των κρατών μελών. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας σχετικά με τις εκτοξεύσεις Ε, τον Αύγουστο για τον Γαλιλαίο. Είναι ένας πολύ περίπλοκος τομέας. Και τα θέματα αυτά και οι διαδικασίες αυτές είναι εξαιρετικά περίπλοκες. Εμείς απογοητευθήκαμε ιδιαίτερος βέβαια για το συμβάν. Ε, κάποιες, κάποια πρώτα συμπεράσματα από το άτυχο αυτό συμβάν δείχνουν ότι οι δορυφόροι μας είναι μεν καλοί, είναι ιδιαίτερα προχωρημένοι και λειτουργούν πάρα πολύ σωστά. Και η δυσλειτουργία προκλήθηκε από το τελευταίο τμήμα του πυράβλου, του εκτοξευτήρα. Και γίνεται μια συνεχής τεχνική έρευνα για το πώς συνέβη το ατύχημα αυτό και πώς θα το αποφύγουμε στο μέλλον. Είμαστε σαφείς σε αυτό. Δεν μπορούμε εμείς ε, να, να συνεχίσουμε με αυτού του είδους ε, τους εκτοξευτές διότι ε, θα πρέπει τα χρήματα και τα χρήματα των φορολογουμένων να μην χρησιμοποιούνται για τέτοιου είδους καταστάσεις. Έχουμε μια ειδική σύμβαση για τα επόμενα δύο χρόνια για τρεις εκτοξεύσεις. Μπορεί να μεταφέρει ο εκτοξευτήρας αυτός με τον οποίο έχουμε συμφωνία ε, τέσσερις δορυφόρους και όχι δύο είναι ευρωπαϊκής ε, σχεδίασης και νομίζω ότι με τους Αριάν, τις εκτοξεύσεις Αριάν θα μπορέσουμε εν πολλής να αντισταθμίσουμε τις καθυστερήσεις που προκλήθηκαν από τις εκτοξεύσεις Άιρους. Τώρα για την γραφειοκρατία. Ε, φυσικά και θα είμαστε απολύτως σοβαροί στην αντιμετώπιση της. Θα χρησιμοποιήσουμε και τα REFIT για να αξιολογήσουμε τις νομοθεσίες οι οποίες θα χρήζουν τροπολόγησης και αλλαγές. Και εφόσον έχετε συγκεκριμένες ιδέες για το ποιες ε, ε, νομοθετικές ρυθμίσεις πρέπει να καλυφθούν εδώ, θα συνεργαστώ μαζί σας όσο στενότερα μπορώ, σεβόμενοι το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ο σας ευχαριστώ. Είμαι εδώ στο βάθος κύριε Σεύκοβιτς. Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας μέχρι τώρα. Θα αναφερθώ στις γραπτές σας απαντήσεις για την αηφορία στις μεταφορές. Είναι απογοητευτικές λίγο γιατί δεν είναι συγκεκριμένες. Γι' αυτό θα σας βοηθήσω να γίνετε πιο συγκεκριμένους. Λοιπόν θα δούμε πώς θα τα πάτε. Δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Πρώτον, ότι στα πλαίσια του πακέτου και των στόχων 2030 δεν υπάρχουν και πάρα πολλά για τις μεταφορές, ενώ η Λευκή Βίβλο ε, φαίνεται ότι θα χρειαζόμαστε για τις μεταφορές συγκεκριμένα ε, μέσα για μετά το 2020, ε, τι θα γίνει με τις οδηγίες οι οποίες θα εκρεμούν μετά το 2020 τώρα για τις αερομεταφορές. Η ΙΚΑΟ θα πρέπει να δώσει προτάσεις για τις παγκόσμιες αερομεταφορές το 2016. Θα πιέσετε προς την κατεύθυνση αυτή, γιατί αν αφήσετε το ΙΚΑΟ μόνο του, τότε δεν θα γίνει απολύτως τίποτα. Σας ευχαριστώ που με βοηθάτε να γίνω πιο συγκεκριμένο στις αξιολογήσεις μου. Και σας ευχαριστώ και για τις ιδέες τις οποίες προτείνατε. Σχετικά τώρα με την κατάσταση μετά το 2020 και σε σχέση με τους στόχους σαν παράδειγμα για τα βιοκαύσιμα. Είστε εμπειρογνώμων σε σχέση με αυτά και γνωρίζετε ότι τα αποτελέσματα με τη χρήση των, ε, πρώτης, των ε, βιοκαυσίμων πρώτης γενεάς δεν ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα λοιπόν ε, με τα εναλλακτικά καύσιμα. Υπάρχουν νέες τεχνολογίες και οι οποίες ελπίζω ότι μετά το 2020 θα βοηθήσουν. Ε, και σε σχέση με τους στόχους της μόλυνσης ε, της ατμόσφαιρας, ιδιαίτερα στις πόλεις μας όπου υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, οι νέες τεχνολογίες και οι νέες μορφές μεταφορών που να είναι καθαρές, που να χρησιμοποιούν τις καινοτόμες τεχνολογίες είναι απαραίτητες και θα πρέπει να είναι και σωστά διατροπικές με την έννοια ότι θα δώσουν κίνητρα στους ε, πολίτες να αφήσουν τα αυτοκίνητά τους στην κατοικία τους. Αυτό θα μειώσει τη μείωση της ατμόσφαιρας ε, και θα απελευθερώσει τους δρόμους. Ε, αυτός είναι ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο θα απαντήσω στο πρώτο κομμάτι της ερώτησής σας. Τώρα, για το ΙΚΑΟ. Ξέρετε ότι η κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ο λίγων περίπλοκη, διότι δεν είμαστε μέλη του ΙΚΑΟ αλλά παρατηρητές. Επαφιέμεθα δηλαδή στην συνεργασία με τα κράτη-μέλη και στο συντονισμό των πολιτικών των κρατών μελών σχετικά με τη διαδικασία λήψης απόφασης στο ΙΚΑΟ. Θα χρησιμοποιήσω όλες τις επαφές τις οποίες έχω στον τομέα των ευρωπαϊκών μεταφορών με τους υπουργούς που θα είμαι σε επαφή έτσι ώστε οι θέσεις ε, του Συμβουλίου να είναι σωστά συντονισμένες. Ένα ερώτημα για τις οδικές μεταφορές και τον ανταγωνισμό στις οδικές μεταφορές. Είναι απαραίτητο στην περίπτωση αυτή <clears throat> να υπάρξει σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας και αυτό δεν θα πρέπει να μείνει μονάχα στα χέρια των κρατών μελών. Είδαμε τους τελευταίους μήνες πολλά προβλήματα και ιδίως σε ό,τι αφορά την ε, διαρρύθμιση για το χρόνο ανάπαυσης και χρόνο οδήγησης. Στη Γαλλία, παραδείγματος χάρη, δεν θα θεωρεί ότι η ανάπαυση στην καμπίνα του φορτηγού είναι πραγματικός χρόνος ανάπαυσης και κινδυνεύουν οι οδηγοί με πρόστιμα 3.000 ε, ευρώ. Ενώ σε άλλες χώρες επιτρέπεται η ανάπαυση στην καμπίνα του φωτιού. Εσείς ως Επίτροπος τι δράση θα αναλάβετε για να αντιμετωπίσετε τα θέματα της εφαρμογής νομοθεσίας αυτού του είδους ώστε να εφαρμόσετε με ισόρροπο τρόπο σε όλες τις χώρες και ακολουθώντας αυτό που είπε ο κύριος Ρικέ, τι θα κάνετε με τη φιλελευθερωποίηση σε επίπεδο καμποτάζου. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Σεύκοβιτς. Πιστεύω ότι όλα τα ερωτήματα τα οποία θέτεται καταδεικνύουν αυτό το οποίο είπα ήδη και εγώ, ότι αυτό που είναι απαραίτητο στις οδικές μεταφορές είναι να υπάρχει μια σε βάθος εξέταση της τωρινής κατάστασης του μεταφορικού τομέα και τις τωρινές κατάστασεις της νομοθεσίας και θα πρέπει να κάνουμε τα εξή. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να διευκρινίσουμε την νομοθεσία αυτή, δεύτερον να την απλοποιήσουμε και τρίτον να εμπλέξουμε τους κοινωνικούς εταίρους για να δούμε πώς θα πρέπει να τροποποιηθούν τα πράγματα και θα πρέπει να συνεργαστούμε μαζί τους ώστε να εξασφαλίσουμε <clears throat> ότι θα μπορέσει να υπάρξει σεβασμός των κοινωνικών τους δικαιωμάτων στον τομέα των μεταφορών και θα έχουν μια κοινή πλατφόρμα για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και φυσικά ό,τι προκύψει από όλα αυτά θα πρέπει να εφαρμοστεί. Η πρακτική αυτή που αναφέρατε για τη Γαλλία για τον χρόνο ανάπαυσης ε, μπορώ να σας πω ότι το ίδιο ισχύει και στο Βέλιο. Δεν έχω δει σε άλλες εθνικές νομοθεσίες μια τέτοια σαφή μορφή περιορισμού ότι δεν μπορεί κανείς να περάσει το χρόνο ανάπαυσης μέσα στην καμπίνα του φωτιού. Προτού όμως καταλήξουμε σε βεβαιασμένα συμπεράσματα, αυτό το οποίο κάνουμε τώρα και που θέλω να συνεχιστεί, είναι να ζητήσουμε διευκρινήσεις από τη Γαλλία και το Βέλγιο μέσω του λεγόμενου πιλότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του συστήματος αυτού που μας επιτρέπει να λύσουμε προβλήματα όταν δεν υπάρχει επακριβής εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα θέσουμε το θέμα αυτό με τις αρχές του Βελγίου και της Γαλλίας και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια θετική λύση η οποία δεν θα είναι διακριτικού χαρακτήρα και θα σέβεται την τωρινή κείμενη νομοθεσία. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Έχω την εξή ερώτηση. Για την κατασκευή δρόμων. Στη χώρα μου έχουν κατασκευαστεί πολλοί δρόμοι. Αλλά με κάποιο παράδοξο τρόπο, δηλαδή γίνονταν διάφορα κομμάτια αυτοκινητοδρόμων χωρίς όμως σύνδεση μεταξύ τους. Κάπου ξαφνικά σταμάταγε ο δρόμος. έργο υποδομών πρέπει να είναι έργο το οποίο παραδίδει αποτέλεσμα 100% λειτουργικό. Λοιπόν, σκοπεύετε να κάνετε κάτι για να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο κατασκευάζονται οι δρόμοι. Να μην γίνεται τμηματικά η κατασκευή. Έτσι ώστε αν δεν είναι ε, ολοκληρωμένος ο δρόμος να μην μπορεί να παραδίδεται. Θα πρέπει να συνδέεται το ένα σημείο, το Α με ένα σημείο Β. Απάντηση. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Πολωνία. Αντίστοιχα προβλήματα έχουμε σε αρκετά κράτη-μέλη. Δεν πιστεύω ότι ήταν εσκεμμένες πάντοτε αυτές οι επιλογές. Μερικές φορές έχουν να κάνουν με την ε, διαδικασία των προμηθειών και ενστάσεις που μπορούν να τραβήξουν επί μακρόν, ε, η ανάγκη για την εξαγωγή μιας πολύ αυστηρής περιβαλλοντικής μελέτης για το συγκεκριμένο έργο. Πάντως συμφωνώ μέσα σας ότι θα πρέπει ε, ιδιαίτερα στο πώς θα κριθεί ένα έργο, δηλαδή το να παραδίδεται ένα έργο το οποίο ε, είναι ε, χρηστικό, ε, πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση. Δεν μπορεί να πηγαίνει δηλαδή κάποιος σε ένα δρόμο και ξαφνικά να τελειώνει ο δρόμος και να μην μπορεί να συνεχίσει με τις ίδιες συνθήκες μεταφοράς την πορεία του, να αλλάζουν δηλαδή οι συνθήκες μεταφοράς. Αυτό θα οδηγήσει σε πολλές ε, συμφορήσεις και πολλά άλλα προβλήματα. Συμφωνώ λοιπόν μαζί σας. Και είναι προφανώς πολύ πιο σημαντικό να εστιμαστούμε στα έργα που έχουν ολοκληρωθεί και βελτιώνουν τις υποδομές σε ολόκληρο το χώρο, έργα τα οποία θα γίνεται κατανοητό και για τον ε, Ευρωπαίο πολίτη ότι βελτιώνουν την κατάσταση στην περιοχή του. Που θα μπορεί να δει ότι έχει καλύτερες μεταφορές στην πόλη του ή στην περιφέρεια του. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να υπάρχει πολύ στενή συνεργασία και με τη Γενική Διεύθυνση ε, Περιφερειακής Πολιτικής, ε, με την DG Move για την πολιτική των μεταφορών της κινητικότητας. Ευχαριστώ πολύ, Ιζαμπέλα Ντεμόντα. Θα ήθελα να επανέλθω στο του καμποτάζ. Εσείς είπατε στην εισαγωγή σας ότι είναι ένα σύστημα χρήσιμο έτσι ώστε να μπορούν να μην κυκλοφορούν κενά ε, τα μεγάλα φορτηγά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει διορθωθεί από τις ε, οδηγίες οι οποίες ισχύουν και οι οποίες δημιουργήσαν ψευδεστήσεις. Αναφερθήκατε και στα θέματα των καινοτομιών οι καινοτομίες σε τέτοια φαινόμενα μπορούν να είναι χρήσιμες. Thank Σας ευχαριστώ. Συμφωνώ πράγματι ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με κάποιο τρόπο. Και ο πρόεδρος της Επιτροπής σας πήρε μέρος ε, σε μια συνάντηση όπου τέθηκε το θέμα των οδηγών φορτηγών ε, όπου προτιμούν, ε, η αστυνομία να τους σταματήσει και να τους βάλει πρόστιμα γιατί οι εργοδότες τους, τους ε, πιέζουν πάρα πολύ να οδηγούν κουρασμένοι και να κινδυνεύουν να είναι κίνδυνος για το κοινό και τον εαυτό τους. Λοιπόν προτιμούν οι οδηγοί των φορτηγών στις διεθνείς μεταφορές, τις οδικές, να τους βάζουν πρόστιμα οι αστυνομικοί. Πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε τους κανόνες θα πρέπει επίσης ε, ε, να καλλιεργήσουμε τον πολιτισμό της, ε, του σεβασμού και της υπακοής των κανόνων. Θα πρέπει οι επιχειρήσεις να σέβονται τους κανόνες οι οποίοι είναι σε ισχύ και να σέβονται γενικά τις ευρωπαϊκές ρυθμίσεις. Σε σχέση με το καμποτάζ είναι ένα ευαίσθητο θέμα φυσικά. Είναι κάτι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει αντιληπτό από το κοινό σαν κάτι το οποίο ε, δημιουργεί θέματα κοινωνικού ντάμπινγκ. Αυτό είναι αλήθεια παρά το γεγονός ότι μόνο του 2% των εμπορευμάτων που μεταφέρονται οδικά ανήκουν στην κατηγορία του καμποτάζ. Πρέπει όμως να αντιμεταπιστεί λόγω των κοινωνικών ανησυχιών, των κοινωνικών προβλημάτων και κυρίως λόγω του ότι εάν το καμποτάζ είναι περιορισμένο ε, όταν παίρνουν κάποια εμπορεύματα εν πάση περιπτώσει στην επιστροφή τους μπορούν να κάνουν μόνο τρεις τάσεις σε επτά ημέρες και αυτός είναι ένας από τους λόγους ε, ε, για τους οποίους το ένα φορτηγό στα τέσσερα κινείται κενό στους αυτοκινητοδρόμους μας. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τα αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά με συνολικό τρόπο και θα πρέπει να καταλήξει σε απλούς κανόνες οι οποίοι να είναι δίκαιοι και οι οποίοι να δείχνουν ότι αντιμετωπίζουμε τα του περιβάλλοντος με υπεύθυνο τρόπο και οι κανόνες θα πρέπει να γίνονται σωστά κατανοητοί και φυσικά σεβαστοί. Μασιμιλιάνο Σαλίνη, σας ευχαριστώ. Κύριε Σεύκοβιτς, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Αναφερθήκατε, λέει ο κύριος Λίνη, για τις σιδηροδρομικές μεταφορές και τη διαχείρισή του στο σύστημα διαχείρισης, το ERTMS. Θα έπρεπε να είναι ενοποιητικός παράγων για τις σιδηροδρομικές μεταφορές θα διευκόλυνε την διαλειτουργικότητα πέρα από τα σύνορα. Σε τεχνικό επίπεδο παραμένουν θέματα σχετικά με τις προδιαγραφές του RTMS. Έχω λοιπόν δύο ερωτήσεις γύρω από αυτό. Η πρώτη, θα συμφωνήσετε ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε τα πρώτα βήματα που θα οδηγήσουν στη σταθεροποίηση του ERTMS και των προδιαγραφών της. Και δεύτερον, θα διασφαλίσετε ότι η Ευρωπαϊκή Σιδηροδρομική Υπηρεσία να είναι υπεύθυνη και για τις δύο πλευρές ε, αδειοδότησης και του υλικού και για το κινητό επίσης υλικό. Σας ευχαριστώ. Υπογραμμίσατε ένα θέμα σημαντικότατο για το μέλλον των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων το σύστημα ERTMS εκτιμάται από όλους τους εμπειρογνώμονες ότι είναι πολύ σύγχρονο ε, και τα σήματα κυκλοφορίας είναι ιδιαίτερα προχωρημένα τεχνικά και αυτή τη στιγμή σε εφαρμοστεί σημαίνει ότι θα έχουμε περισσότερα τρένα ε, στα δίκτυα, περισσότερους επιβάτες, περισσότερα ε, εμπορεύματα και περισσότερη ασφάλεια. Βέβαια η ανάπτυξη του συστήματος αυτού ε, είναι κάτι το οποίο τώρα ολοκληρώνεται και θα θέλαμε να μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε γρηγορότερα από ό,τι προβλέπεται. Για να το πετύχουμε αυτό, η λύση στο πρόβλημα αυτό είναι να υπάρξει ένα σωστό διαχειριστικό σύστημα για την εφαρμογή του συστήματος και να πιέσουμε για την εφαρμογή του συστήματος αυτού στα κεντρικά σιδηροδρομικά ευρωπαϊκά δίκτυα, εκεί όπου χρειάζεται κυρίως περισσότερο ε, από ε, αλλού. Το σύστημα λοιπόν αυτό, αν ε, ίσχυε κάποια από τα τραχικά ατυχήματα που είχαμε τον προηγούμενο χρόνο θα είχαν αποφευθεί, γιατί το σύστημα είναι καλύτερο και ασφαλέστερο. Η υπηρεσία αυτή θα πρέπει να είναι λοιπόν και για το κινούμενο υλικό, για τα βαγόνια δηλαδή και για το δίκτυο και για την σωστή εφαρμογή ε, του συστήματος ERTMS. Θα ήθελα επίσης να πάω ένα βήμα παραπέρα και να πω ότι θα έπρεπε ίσως να είναι ε, και υπεύθυνη για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις τεχνικές προδιαγραφές των ανταλλακτικών των, ε, ε, των οχημάτων των συνδυοδρομικών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μας είπατε ότι έχετε εργαστεί σε μια απλή εργασία και όλοι χαιρόμαστε για το γεγονός ότι ξέρετε τι θα πει να ζει κανείς με περιορισμένα ορισμένες αποδοχές. Ήμουνα οδηγός φορτηγού για 30 χρόνια και έχω γυρίσει όλη την Ευρώπη. Στο παρελθόν δεν υπήρχαν τόσα άδεια φορτηγά, υπήρχε περισσότερο καμποτάζ, αλλά με το νέο σύστημα κανόνων που ισχύει έχουμε ανοίξει τις πόρτες στους κακούς μέσα σε εισαγωγικά, αυτούς που φοράνε τα μαύρα καπέλα στα έργα. Έχουμε ένα πρόβλημα με τις ε, ε, πλαστές άδειες οδήγησης για τα φορτηγά. Από το ίντερνετ για 400 ευρώ μπορεί κανείς να αγοράσει ένα διαβατήριο, ένα δίπλωμα οδήγηση επαγγελματικό και όλη την τεκμηρίωση. Μπορεί ένα άτομο να έχει τρία τέτοια διπλώματα και να οδηγεί 24 ώρες το 24 γιατί δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Αστυνομία που να μπορεί να ελέγξει τη γνησιμότητα αυτών των αδειών οδήγηση. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο αυξάνεται. Είναι ένας διεθνής κίνδυνος. Οι διαμεθοριακές μεταφορές είναι πολύ σημαντικές. Αλλά πλήττονται από αυτό το πρόβλημα. Ένας κανονικός ε, οδηγός θα πρέπει να καταγραφεί στην τοπική αστυνομία της περιοχής του. Αν όμως η εθνική αστυνομία έχει τη δυνατότητα να ελέγξει ότι είναι πράγματι ε, νόμιμη και όχι πλαστή η άδειά του, αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν ήταν ερώτημα αυτό, λέει ο κύριος Σεύκοβιτς. Ή μια δήλωση. Πιστεύω ότι δεν ήταν και η πρόθεσή σας γιατί ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η δουλειά <clears throat> των οδηγών φορτηγών και εγώ δεν θεωρώ ότι οι οδηγοί οι οποίοι δεν κάνουν καμποτάζ είναι οι κακοί στο επάγγελμα αυτό. Κάνουν διεθνεί μεταφορές και γυρίζουν και πάλι στην βάση τους και προσπαθούν να βρουν κάποιο φορτίο στην επιστροφή ώστε να μην κυκλοφορεί το φορτηγό τους άδειο. Αν τώρα υπάρχουν καταχρήσεις του συστήματος, συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Αλλά το ερώτημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εδώ το έχω τονίσει και πάλι είμαι έτοιμο να απλοποιήσω και να διευκρινίσω του κανόνε ώστε να υπάρχει σωστή εφαρμογή του. Αλλά η αστυνόμευση των κανόνων αυτών θα πρέπει να γίνει από τι εθνικέ αρχέ γιατί αυτοί έχουν το δικαίωμα να το πράξουν. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ρωτήσω για περιοχές με ειδικά χαρακτηριστικά, ορεινές, παράκτιες, περιοχές που χρειάζονται δηλαδή επενδύσεις λόγω των ιδιαίτερων οικονομικών συνθήκων, αλλά και που έχουν ιδιαίτερα οικολογικά χαρακτηριστικά. Εγώ εκπροσωπώ την ε, Ουαλία, στην οποία δεν προβλέπονται διάδρομοι των Τσέντσι. Έχουμε ωστόσο ταυτόχρονα ανάγκη για καλές ε, διασυνδέσεις ε, σιδηροδρομικές. Είπατε ότι οι μεταφορές αφορούν τους πάντες. Ταυτόχρονα όμως μπορεί και να αποκλείουν κάποιους πολίτες. Πώς μπορείτε λοιπόν να εξασφαλίσετε ότι ε, επενδύσεις και υποστήριξη ορθές και σκόπιμες εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα για τις περιοχές με σεβασμό βέβαια και προς τον τουρισμό και τις περιοχές αυτές. Ευχαριστώ πολύ και βέβαια είναι ένα πολύ σημαντικό όσο και δύσκολο, δυσεπίλητο ζήτημα. Αντιλαμβάνομαι την ε, οπτική σας. Οι μεταφορές είναι πολύ σημαντικές όχι μόνο ως παράγον συμπερίληψης, ενσωμάτωσης, ολοκλήρωσης οικονομίας, συμπερίληψης των, των ε, πόλεων στις περιφερειές τους σε εθνικό αλλά και διεθνές δίκτυο. Ταυτόχρονα όμως, εάν κοιτάξουμε τις ευρωπαϊκές πολιτικές και τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό κυρίως δυστυχώς, δεν αρκεί για να καλύψει όλες τις ανάγκες. Ελήφθη μια απόφαση λοιπόν ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα διευρωπαϊκά δίκτυα και κυρίως σε μια συμφόρηση στους τομείς όπου προξενούνται σημαντικά προβλήματα με επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη και τα σημεία όπου λείπουν οι σύνδεσμοι. Για την περίπτωση της Ουαλίας συγκεκριμένα που ρωτήσατε. Βεβαίως, εάν δεν έχει ενταχθεί στο σύστημα των διευρωπαϊκών δικτύων των μεταφορών θα είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί μια λύση για την Ουαλία λόγω ακριβώς των κανόνων που έχουν υιοθετηθεί, γιατί αυτοί ε, στοχεύουν ειδικά στην ε, αξιοποίηση κονδυλίων για τις προτεραιότητες των διευρωπαϊκών δικτύων. Ευχαριστώ κύριε Σμαρτέζα. Κύριε υποψήφιε ε, πίτροπε, δεν απαντήσατε σε μία ερώτηση της κυρίας Ντέλη των Πρασίνων σχετικά με τη σύνδεση της γραμμής σιδηροδρομικής υψηλής ταχύτητας Λιών-Τωρίνου. Είναι σκανδαλώδες ε, να ξοδεύονται ε, δημόσια χρήματα για τέτοιου είδους ε, επενδύσεις. Είχε αποφασίσει έτσι και αλλιώς η Ιταλική κυβέρνηση να μειώσει κατά το 1 τρίτο τη συγχρηματοδότηση την εθνική. Το κόστος από ό,τι φαίνεται όμως του έργου αυτού συνεχίζει να αυξάνεται. Η οικονομική κατάσταση στην Ιταλία και την Γαλλία σίγουρα δεν έχει βελτιωθεί και οι ανησυχίες για την αηφορία, την οικονομική και την ε, ε, οικολογική ε, δυστυχώς αυξάνονται. Μήπως θα έπρεπε λοιπόν εσείς το σύνολο του σχεδίου αυτού να το περάσετε από μια νέα οικονομική εξέλιξη, εξέταση συγγνώμη, ε, ή τουλάχιστον να δώσετε την ανάλυση αυτή σε έναν ανεξάρτητο μηχανισμό και να μην δαπανίσετε περαιτέρω κοινοτικά χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε άλλους τομείς πολύ πιο απαραίτητους για την κοινοτικότητα της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Από ό,τι καταλαβαίνω είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε και στην Ιταλία και στη Γαλλία όπως επίσης και σε ε, ε, φόρα όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να πω εδώ ότι ε, το πρόγραμμα αυτό έχει εγκριθεί. Ο κοινοτικός κανόνας λέει ότι πρέπει να σεβαστώ την απόφαση αυτή. Αυτό το οποίο μπορώ να σας υποσχεθώ είναι ότι σχετικά με την κατασκευή της υποδομής αυτής θα πρέπει να σεβαστούμε και άλλα, άλλες πλευρές και άλλα τμήματα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Να υπάρξει σωστή διαβούλευση με το κοινό. Οι περιβαλλοντικοί κανόνες να γίνονται σεβαστοί. Όλες δηλαδή οι πλευρές αυτές θα καταλήξουν στην τελική έγκριση ενός τέτοιου σχεδίου, ενός τέτοιου προγράμματος. Πρέπει να γίνονται σεβαστοί λοιπόν όλοι οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Τώρα, αν αρχίσουμε να τα συζητάμε όλα αυτά εκ νέου, φοβάμαι ότι θα ανοίξουμε το κουτί της πανδώρας και δεν θα μπορέσουμε να το κλείσουμε στη συνέχεια. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι αυτό το οποίο αποφασίστηκε από το Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο και θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στην εφαρμογή της αποφάσεως αυτής σεβόμενη όλες τις πλευρές της κοινοτικής νομοθεσίας και σεβόμενη όλες τις ρυθμίσεις οι οποίες θα πρέπει ακριβώς όπως είπα να γίνουν σεβαστές. Τελίτσκα να υποστηρίξω αυτά τα οποία είπατε κύριε υποψήφιε επίτροπε σε σχέση με την εφαρμογή της αρχής use it or lose it. Αν δεν τα χρησιμοποιήσεις θα τα χάσεις. Ε, ήδη τέθηκαν ερωτήσεις για τα διόδια στην Γερμανία. Νομίζω ότι ε, το συζητάμε το θέμα αυτό εδώ και 25 χρόνια για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών και δεν το έχουμε πετύχει ακόμα αυτό. Και δεν έχω καταλάβει αν θα ξεκινήσετε εσείς την συζήτηση ε, για το κόστος αυτό το επιπλέον στις μεταφορές. Και όταν αναφέρεστε στον σεβασμό και ε, στην έλλειψη διακρίσεων, Ξέρουμε ότι οι δηλώσεις οι οποίες γίνονται στην Γερμανία κατά κάποιο τρόπο ε, τεκμηριώνουν το επιπλέον αυτό κόστος. Ε, αλλά δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση αυτό ε, να χρησιμοποιηθεί σαν αντιστάθμισμα για το κόστος των εσωτερικών μεταφορέων. Δεν έχω πρόβλημα με τα διόδια δηλαδή, με τα τέλη των διοδίων, αλλά η χρήση τους, σε πάση περιπτώσει, είναι αυτό το οποίο είναι πρόβλημα γιατί όταν αυξάνει κανείς ε, ε, τις γραφειοκρατικές και τις οικονομικές επιβαρύνσεις ταυτόχρονα θα παίρνει και μέτρα ελάφρυνσής τους. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ. Και σίγουρο. ότι μπορώ να υπολογίζω στην υποστήριξή σας για μια πολύ αυστηρή επαλήθευση της στήρησης του κανόνα use it or lose it, αξιοποίησε ή χάνει την ευκαιρία σε αυτό θα είμαστε πάρα πολύ αυστηροί γιατί είναι πολύ περιορισμένοι οι δημοσιονομικοί πόροι. Και το, η δουλειά που έχουμε μπροστά μας είναι πολύ σημαντικά, έχουμε, σημαντική, έχουμε πάρα πολλά μεγάλα έργα και θα πρέπει να αποδείξουμε και να πείσουμε τα κράτη-μέλη ότι θα αξιοποιούν τους πόρους εγκαίρως ή θα κινδυνεύουν να τους χάσουν. Και βεβαίως εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να εφαρμόζονται οι κανόνες αυτοί για δε την κατάσταση τη σχετική με τα διόδια στη Γερμανία. Όπως είπα, αφενός μεν χαίρομαι που ξεκινάει, που ανοίγει η συζήτηση στη Γερμανία. Ο, η αναζήτηση δηλαδή της ε, εσωτερήκευσης εξωτερικού κόστους, γιατί η Γερμανία έχει την τεράστια υποδομή ως χώρα. Ταυτόχρονα όμως βλέπουμε και να κλείνουν γέφυρες και να μην υπάρχει σωστή συντήρηση ορισμένων αυτοκινητοδρόμων. Χαίρομαι λοιπόν που η συζήτηση αυτή άρχισε συζήτηση η οποία αφορά και το πώς μπορεί να εσωτερικευθεί το εξωτερικό κόστος της ε, χρήσης των ε, οδικών υποδομών. Όπως είπα, έχει τεράστια σημασία για μένα η αρχή ο πληρώνει και η αρχή της απαγορεύσεων διακρίσεων. Αυτό θα είναι σαφέστατο εκ μέρους μου, θα καθίσατε σαφέστατο όταν βλέπω, όταν δω συγκεκριμένα το διατακτικό του νόμου που πρόκειται να καταθέσει η γερμανική κυβέρνηση, θα το εξετάσω με απόλυτη αυστηρότητα. Ευχαριστώ, Ρόμπερτ Σίλε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σεύκοβιτς, για τις ε, απαντήσεις σας. Θα ήθελα να επισημάνω ότι με χαρά λαμβάνω το λόγο μετά τον συνάδελφο ο οποίος είχε ε, το συντονισμό του προγράμματος για τη Βαλτική. Θα περιμένετε, φαντάζομαι, θα αναμένετε αρκετή υποστήριξη από την Επιτροπή μας ε, για το θέμα της Βαλτικής. Εμείς έχουμε μια ισχυρή βρετανική στηρητική ε, ομάδα στην ε, ομάδα των στηρητικών μεταρρυθμιστών που όμως απουσιάζει αυτή τη στιγμή εκπροσωπός της διότι βρίσκεται σε μια ε, διάσκεψη στην Βρετανία σε ένα συνέδριο, αλλά έχω αναλάβει εγώ να τον εκπροσωπήσω. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω για την πρωτοβουλία για τους ενιαίους ευρωπαϊκούς εθέρες που μπορεί να παρεμποδιστεί από διάφορα μέτρα ε, που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη. Πώς μπορούν λοιπόν να επιταχυνθούν αυτές οι πρωτοβουλίες. Νομίζω ότι είχατε και την πιο εύκολη ερώτηση εγώ να υποβάλω. Ευχαριστώ. Ναι, ναι, ναι και σας ευχαριστώ θερμά. Για την ερώτηση λοιπόν αυτή. όποιος θέλει να προωθήσει ένα αίσιο μέλλον, ένα καλό, μια καλή προοπτική για τους ευρωπαϊκούς εθέρες, θα πρέπει να αισθάνεται μια κάποια δυσφορία για το ότι δεν έχουμε προχωρήσει αρκετά. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση με τα λεγόμενα FABS, την ε, εξασφάλιση εννέα εδαφικών στοιχείων, που χωρίς να είναι ιδεώδης λύση γεννούν νέες και ποικίλε ευκαιρίες για πιο σύντομους δρόμους, για πιο, σύντομες δηλαδή για εξοικονόμηση χρόνου, πόρων, εκπομπών στις αεροπορικές πτήσεις. Όπως είπα, αυτό ισοδυναμεί σε 5 δισεκατομμύρια ευρώ κατέτος. Όπως είπα, Μέχρι τώρα η πρόοδος είναι μάλλον περιορισμένη και αισθανόμαστε μια κάποια απογοήτευση. Θα προτείνω λοιπόν καταρχάς να αξιοποιηθούν περισσότερο τα κριτήρια αποτελεσματικότητας ή απόδοσης καλύτερα, όπου θα πρότεινα στα FAPS να ε, προσμετράτε ε, το κριτήριο της απόδοσης και πόσο θα μπορούσε ακόμη να συντομεύσει μια πτήση, να περιοριστούν οι εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα, να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της πτήσης μέσα σε ένα ΦΑΠ που θα είναι συγκρίσιμο με το ΦΑΠ κάποιου άλλου και έτσι μπορούμε να ξεκινήσουμε ένα υγιή ανταγωνισμό που θα δείχνει πώς ένα ΦΑΠ έχει καλύτερα αποτελέσματα από κάποιο άλλο και πόσα χρήματα χάνονται κάπου αλλού. Και βεβαίως Εάν δούμε ότι ε, υπάρχει μια συνεχιζόμενη ε, ε, παραγνώριση των αρχών των ΦΑΠΣ, τότε θα πρέπει να διαρχίσουν και διαδικασίες επιπαραβέας. Διότι δεν μπορούμε να αφήσουμε να χάσουμε περισσότερο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ουιέλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Σεύκοβιτς, είμαι εδώ αμέσως μπροστά σας. Ως ε, ο τελευταίος ομιλητής από τους σοσιαλιστές και αντιπρόεδρος της Επιτροπής αυτής θα ήθελα να σας τονίσω ότι μετά από σχεδόν τρεις ώρες, μια μαραθώνια ακρόαση, ξέραμε ότι ήσασταν εξαιρετικός διπλωμάτης, το είδαμε από το βιογραφικό σας, αλλά είσαστε και πάρα πολύ καλά προετοιμασμένος για τα θέματα μεταφορών και δείχνετε σημαντικό ενθουσιασμό για τα θέματα αυτά. Είδα την ε, γραπτή σας απάντηση και είχα κάποια ερωτήματα αλλά τα έχετε απαντήσει όλα. Μπορείτε λοιπόν να χαλαρώσετε, ας αφήσουμε τις μεταφορές και πέστε μου το εξή Τα επόμενα χρόνια ως ένας γείτονας από την κεντροανατολική Ευρώπη με την ιστορία της χώρας σας. πώς, θα είναι, πώς είναι το μέλλον της ε, Ευρώπης σε επίπεδο μεταφορών. Τι μπορούμε να κάνουμε που είναι το πιο σημαντικό για τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ και για την πιο φιλοσοφικού χαρακτήρα αυτή η ερώτηση. Νομίζω ότι το μέλλον είναι λαμπρό, είμαι αισιόδοξο από αυτή την άποψη. Τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν πολύ δύσκολη εποχή βρεθήκαμε στο χείλος της κατάρρευσης ουσιαστικά της διαδικασίας ευρωπαϊκής ε, ολοκλήρωσης. Αλλά όταν συζητάμε για το πού βρισκόμασταν πριν από 25 χρόνια πριν και πού βρισκόμαστε τώρα, είναι η ιστορική η πρόοδος που έχουμε επιτύχει και παρά τα τελευταία χρόνια της κρίσης δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα πόσο έχει αλλάξει η Ευρώπη και πόσο έχουμε προχωρήσει και πόσο πολύ πρέπει να αξιολογήσουμε θετικά τα θέματα αυτά. Εγώ μεγάλωσα στην Πρατισλάβα πίσω από το συνδρόμου παραπέτασμα. Νόμιζα όταν ήμουν νέο ότι ποτέ δεν θα μπορούσα να φτάσω στην Αυστρία, θα με σταματούσαν στα σύνορα. Είναι ένα θαύμα αυτό που έχει συμβεί και πρέπει να το ομολογήσω. Το καταπληκτικό είναι τα παιδιά μας το παίρνουν για δεδομένο. <clears throat> Θεωρούν δεδομένο ότι δεν υπάρχουν σύνορα. Δεν υπάρχουν συνοριακοί έλεγχοι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι αυτό το οποίο θα έπρεπε να συμβαίνει. Πρέπει και εμείς για τις μεταφορές να κάνουμε το ίδιο. Πιστεύω ότι αυτή η Επιτροπή, η Επιτροπή σας είναι ιδιαίτερα δεσμευμένη και προσφελωμένη να γίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν πάρα πολλοί εμπειρογνώμονες στην Επιτροπή αυτή που έχουν περάσει όλη τους την καριέρα στον τομέα των μεταφορών. Έχω συναντήσει πολλούς από εσά και ξέρω πόσο υποστηρίζετε την Ευρώπη και πόσο θέλετε να εργαστείτε για να μπορούμε να έχουμε πραγματικά ένα ε, ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο, χωρίς σύνορα, χωρίς ελέγχους, χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς προστατευτισμό, μία μονάχα ενιαία Ευρώπη μεταφορών. Υπάρχει όμω και μια ακόμα ερώτηση παρά τα χειροκροτήματα. Η κυρία Λουκατσιεύσκα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Ε, περνάω κατευθείαν στην ερώτησή μου και ότι ο υποψήφιος επίτροπος έχει απαντήσει σε μεγάλο βαθμό σε αυτό που θέλω να ρωτήσω. Θα τη θέσω. Πώς αξιολογείται την κατάσταση τώρα για το καμποτάζ ε, όπως αυτή επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι θα πρέπει να πράξουμε προκειμένου να βελτιώσουμε τις οδικές μεταφορές, να ε, ενισχύσουμε το δυναμικό τους την παραγωγικότητά τους και τι πρέπει να κάνουμε για να ε, εφαρμοστούν επιτέλους οι διατάξεις οι οποίες δεν βρίσκονται ακόμη ενισχύ. Πιστεύω ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βρει έναν τρόπο να βοηθήσει τους ε, οδικούς μεταφορείς ε, που δεν έχουν ακόμα μπορέσει να λύσουν το πρόβλημα της διαμετακόμισης λόγω του εμπάργου που επιβάλλονται σε ορισμένα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατευθύνονται προς τη Ρωσία. Ευχαριστώ. Απάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Το θέμα της διαμετακόμισης είναι προφανώς πολύ ε, λεπτό, έχει πολλές ε, συνέπειες και σε κοινωνικό επίπεδο, καθώς πολύ μεγάλο τμήμα των μεταφορών μας περνάει μέσα από αυτό. Πρέπει να απλουστεύσουμε και να διευκρινίσουμε τους κανόνες, νομίζω. Διότι Πρέπει πάνω απ' όλα να αποκαταστήσουμε το αίσθημα της κοινωνικής ασφάλειας για τον οδηγό του φορτηγού. Πρέπει και είναι πολύ σημαντικό και εδώ θα πρέπει να κληθούν και οι εθνικές αρχές να ενισχυθεί η επιβολή, η εφαρμογή των κανόνων που ισχύουν. Η τεχνολογία επίσης, η παραδείγματι, στο, στις μετρήσεις. Ο υπολογισμός ε, του εάν τηρούνται οι κανόνες, ο ψηφιακός ταχογράφος, οι νέες τεχνολογίες οι οποίες και χάρη στο νέο σύστημα, στα νέα συστήματα πλοήγησης και το δυναμικό που προσφέρουν οι δορυφόροι ε, στην Ευρώπη μπορεί να είναι ένα ζήτημα αξιολόγηση. Και όταν η Ευρώπη έχει το, την πρώτη θέση, την πρωτορική θέση στην επιμελητία, τότε μπορούμε να βοηθήσουμε και τα κράτη-μέλη να σχεδιάσουν καλύτερα το ε, χρόνο οδήγηση την διαχείριση του φορτίου, την επιμελητιακή ολοκλήρωση σε ένα διατροπικό είδος μεταφορών σε ένα χώρο μεταφορών που οικοδομούμε στην Ευρώπη. Όπως είπα, ένα στα τέσσερα φορτηγά κυκλοφορεί κενό φορτίου. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να λύσουμε. Για δε τα προϊόντα που εξάγονται προς τη Ρωσία είναι απαράδεκτη κατάσταση που έχει επέλθει με το εμπάργκο. Στο προσεχές ε, στην προσεχή συνεδρία της Επιτροπής θα το συζητήσουμε πάρα πολύ σοβαρά. Θα βρούμε μια λύση συνεργασία με τις ρωσικές αρχές γιατί δεν είναι δυνατόν να υποφέρουν οι οδηγοί των φορτηγών μας επειδή υπάρχουν εντάξει.